Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σήμερα το απόγευμα, με ιδιαίτερη χαρά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάρκα Σπρέγκερ, που είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Νοσημάτων. Είναι εδώ και όπω έρχεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ήρθε να μα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού αυτού Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και να σημειώσω τις δικές σας ανησυχίες αλλά και παροτρύνσεις. Χαίρομαι που επίσης μου είπατε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφάνειες. Και γιατί το κάνω αυτό, γιατί μου είπατε ότι θέλετε να είμαι πιο ανοιχτό όσον αφορά τα αποτελέσματα που έχουμε από τα διάφορα κράτη-μέλη όταν πρόκειται για τις μεταδοτικέ ασθένειε. Θα σας δώσω λοιπόν στοιχεία. Η παρουσίασή μου αποτελείται από τρίτηματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας και τέλος θα σας μιλήσω για τα συμπεράσματα και τις ε, συνέπειες της πολιτικής μας. Κοιτάξτε την πρώτη μου διαφάνεια. Η πρώτη μου διαφάνεια έχει να κάνει με τις κοινοποίησεις που έχουμε όσον αφορά την εφηματίωση για 100.000, ε, μάλλον. Έχουμε εδώ πέρα, βλέπετε στη Ρωσία, ένα μεγάλο αριθμό. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν τα πάνε καλά. Αυτές που φαίνονται σε κόκκινο. Βλέπετε ότι είναι η Ρουμανία, για παράδειγμα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τίθεται το ερώτημα τι γίνεται στη Ρουμανία. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ότι οι χώρες που βρίσκονται σε πιο καλή κατάσταση είναι χώρες στις οποίες υπάρχει επιπολασμός. Τώρα, ποιο είναι το άσχημο νέο σε όλα αυτά. Το άσχημο νέο είναι ότι υπάρχουν ε, πολλές αντιστάσεις στα φάρμακα. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα και για τους ασθενείς, αλλά και για την κοινωνία, γιατί η θεραπεία είναι πολύ ακριβή και δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα για τους ίδιους τους ασθενείς. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα δράσης για την φυματίωση με στόχο καλύτερη διάγνωση όσον αφορά τις περιπτώσεις που αντιστέκονται στα αντιβιωτικά και στα φάρμακα ε, για την ασθένεια αυτή. Ε, προσπαθήσαμε δηλαδή να βοηθήσουμε ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα ασφάλισης, ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση της φυματίωσης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό βλέπετε, γιατί αν μπορέσετε να διαγνώσετε σε ένα αρχικό στάδιο την ασθένεια, είναι καλό για τον ασθενή πρώτα απ' όλα, γιατί έτσι ο ασθενής ε, αντιστέκεται καλύτερα. Είναι καλό για την κοινωνία, διότι δεν θα μεταδοθεί η ασθένεια και θα εξαφανιστεί μετά από λίγο καιρό. Εδώ τώρα υπάρχει βέβαια και κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ ελκυστικό, όπως είναι η θέρμανση του κλίματος ή ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της βιοπικιλότητας, όμως για τους ευάλωτους ανθρώπους, τους πιο φτωχούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο αριθμός των ε, διαγνώσεων που έχουμε για το AIDS. Το 2008 για παράδειγμα. Βλέπετε και εδώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ κυρία Ρότα Τάκμαρ Βέρεντ. Γιατί εσείς ζητήσατε να είμαστε πιο ανοιχτοί. Ενά, Λοιπόν, είμαστε πιο ανοιχτοί και μπορούμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αναχώρα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορές. Όμως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί διαδίδεται το έτσι στην Ευρώπη. Γιατί διαδίδεται μεταξύ ανδρών που έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Υπάρχει αύξηση της παρουσίας του AIDS σε αυτήν την κατηγορία. Υπάρχουν βέβαια μεγάλες διαφορές. Πριν από ένα χρόνο, το άτομο επαφής που έχουμε, η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκης, ε, φιλοξένησε ένα επιστημονικό σεμινάριο και την ε, 1 Δεκεμβρίου έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για το AIDS. Πάλι η Μαρίνα θα φροντίσει γι' αυτό. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η μέρα. Γιατί θα ξεκινήσουν οι πρώτες επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά ε, τα, τις εξετάσεις AIDS. 30% των ατόμων που έχουν AIDS δεν γνωρίζουν ότι έχουν τον ιό. Αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι δεν ε, ακολουθούν καμία θεραπεία και ότι μπορούν να ε, μεταδώσουν την ασθένεια και σε άλλους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και εδώ η διάγνωση να γίνεται έγκαιρα. Και εδώ υπάρχει από τη δικιά μας την πλευρά μια προσθέμενη αξία ότι φροντίζουμε γι' αυτό. Μια άλλη περίπτωση, πατήτιδα Β και Γ. Ίσως να μην είσαστε τόσο εξοικειωμένοι με τις ασθένειες αυτές και να σας ακούγονται πολύ εξωτικές, αλλά σας προφορώ ότι η πατήτιδα Β και Γ είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους καταλήγει κανείς να έχει καρκίνο του ύπατος. Και εδώ υπάρχουν διαφορές. Πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας και δείξαμε ότι δεν κάνουν έλεγχο στις έγκυες γυναίκες για τις ασθένειες αυτές όλες οι χώρες. Προγενετικό έλεγχο δηλαδή. Αν γίνει προγενετικός έλεγχος, το βλέπεις και δίνεις και τα σωστά φάρμακα, γράφεις τη σωστή θεραπεία. Αν όμως δεν το ξέρει η μητέρα, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια στο παιδί της. Με ξέπληξε πάρα πολύ η ομιλία της, του κύριου Πίτελη στην διάσκεψη που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Όμως χρειάζεται και πολιτικά να δοθεί σημασία στις ασθένειες αυτές. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη ασθένεια. Η μαλάρια. Ναι, έχει εξαφανιστεί σε ένα βαθμό. Βέβαια, αν πας σε μια χώρα που μπορεί να κινδυνεύεις από μαλάρια, παίρνεις χάπια. Όμως πριν από μερικές δεκαετίες είχαμε ε, στην Ευρώπη μαλάρια εξαιτίας ενός ε, κουνουπιού και ήρθαν διάφοροι ειδικοί που ξέρουν τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κουνούπια. Ίσως κάποιος από την Ελλάδα να είναι εδώ. Είναι εδώ κάποιος από την Ελλάδα. Μεταξύ του ακροτηρίου έχουμε εδώ κανέναν ε, Έλληνα. Στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει ο μιλητής, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εμφανίστηκαν τέτοια κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Πολλά. Πάνω από 50 επιβεβαιωμένα κρούσματα. 70% των περιπτώσεων αυτών ήταν άτομα που ασθένησαν σοβαρά. Και 30 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Πράγμα που σημαίνει ότι για αυτή την περιοχή είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή η ασθένεια. Σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί όχι, αλλά αν ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο ιός αυτός επηρεάζει και τον τουρισμό στην περιοχή. Μας ρώτησαν λοιπόν, μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση και να δείτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Τι κάνουμε λοιπόν. Βρήκαμε εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη, δεν είναι και πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν ε, κάποιοι στη Ρουμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, γιατί και από εκεί έχει περάσει η ασθένεια αυτή. Συναντηθήκαμε λοιπόν όλοι μαζί και συναντηθήκαμε και με τους ειδικού από την Ελλάδα. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση αυτή. Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μα. Δεν ξέρω εδώ αν εσεί αναγνωρίζετε όλα αυτά τα είδη κουνουπιών. Πάντως αυτό που είναι πάνω δεξιά είναι εκείνο το οποίο προκαλεί τον ιό και μεταδίδει μάλλον τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ε, μέσα από τα πουλιά ε, μεταφέρεται αυτός ο ιός και όμως απ' Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που διάφοροι εμπειρογνώμονες συναντήθηκαν στην Ελλάδα. Ε, κτηνίατροι και άλλοι ειδικοί από διάφορους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Τι κάνουμε λοιπόν. Να, εδώ βλέπετε τους δικούς μας εμπειρογνώμονες. Να, τρεις. Συζητάμε λοιπόν τις βέλτιστες πρακτικές για να ελέγχονται τέτοιου είδους ασθένειες. Μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια πρώτη περίπτωση ελονοσίας στην Ισπανία. Δεν επρόκειτο για εισαγωγή, δεν ήταν κάποιος τουρίστας δηλαδή, όχι, ήταν κάποιος ντόπιο. Φυσικά και ανησυχήσαμε και οι ισπανικές αρχές ε, ανησύχησαν. Οπότε και πάλι προσπαθήσαμε να δούμε πού οφείλεται. Έχει να κάνει με τις κλιματικές αλλαγές. Πάντως πρόκειται για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων μεταδίδονται οι ασθένειες αυτές. Τώρα εδώ βλέπετε αυτή τη διαφήμιση για τα αντιβιωτικά. Πολλά αντιβιωτικά πρέπει να ξέρετε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πιάνουν. Δεν πιάνουν έτσι κι αλλιώς τα αντιβιωτικά αν έχετε μια ασθένεια που οφείλεται σε ιό. Όμως σε σοβαρές περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς δεν πιάνουν γιατί οι ασθενείς, οι γιατροί πάρα πολύ συχνά ε, γράφουν στους ασθενείς αντιβιωτικά και έτσι έχουν συνηθίσει οι οργανισμοί μας και δεν αντιδρούν. Είχαμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ημέρα ενημέρωσης κατά των αντιβιωτικών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ημερίδες διότι βοηθούν να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. 16 Νοεμβρίου θα έχουμε την τρίτη τέτοια ημέρα ενημέρωσης κατά των αντιβιωτικών. Και χαίρομαι που πάνω από 36 χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή και χώρες δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα φροντίσουν να έχουν την ίδια μέρα και εκείνη σαν μέρα κατά των αντιβιωτικών. Να λοιπόν που η πολιτική ε, στήριξη έχει μεγάλη σημασία. Χρειάζονται και εκστρατείες ενημέρωσης σε όλες τις χώρες. Τώρα, προσπαθώ να φτάσω εδώ στη σωστή εικόνα. Α, ναι, αυτή ήταν που θέλω να σας δείξω. Εδώ, κάθε πρωί στις 11.30 έχουμε συνάντηση μεταξύ μας και συζητάμε τα πάντα. Δηλαδή τι νέα έχουμε επίσημα, τι μας φτάνει από δημοσιογραφικές πηγές, τι μαθαίνουμε και έχει μεγάλη σημασία γιατί έτσι ξεκινάει η αξιολόγηση μιας απειλής. Σήμερα το πρωί φυσικά δεν ήμουνα σε αυτή τη συνεδρίαση, αφού βρίσκομαι εδώ, αλλά ήρθα σε επαφή μαζί τους και σήμερα το πρωί τι μάθαμε, ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις του σκαθαριού αυτού, ένα βακτηρίδιο που προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο. Που προκαλεί δηλαδή εδώ νοσοκομιακές λοιμώξεις. Στην Κίνα, στη Μαλαισία, στο Ισραήλ και σε μερικές άλλες χώρες έχουμε τέτοια εμφάνιση με μεγάλη ένταση. Είναι ένα σούπερ λοιπόν βακτηρίδιο το οποίο διαδίδεται και που τα κοινά, τα συνήθεια αντιβιωτικά δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Πρέπει να βρούμε άλλα, καινούργια αντιβιωτικά. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε επίσης και άλλα θλιβερά νέα, τα νέα της ΑΙΤΙΣ, για τη χολέρα εκεί. Ίσως όλα αυτά να σας φαίνονται υπερβολές. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην ΑΙΤΙΣ θα μου πείτε. Δεν είναι στην Ευρώπη στο κάτω-κάτω. Ναι, αλλά ξέρετε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες τα Χριστούγεννα θα πάνε στην άλλη μεριά του νησιού που βρίσκεται η Αιτή Θα επισκεφθούν δηλαδή την Δομινικανική Δημοκρατία. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αίτη, γιατί οι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται εκεί δίπλα. Και θα μπορούσε κάλλιστα η χολέρα να περάσει και από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση και να είμαστε ενημερωμένοι για να μπορούμε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε επαφές με τους ειδικού στην ΑΕΤ για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έρχομαι λοιπόν τώρα εδώ στην ακρόαση του Απριλίου, όπου σας είχα πει ότι θα έδινα περισσότερη σημασία στην ε, συμφωνία για την έδρα, seat agreement, με τον ε, Σουηδό Υπουργό Υγείας, ότι θα προείδρευα και ότι όντως υπεγράφει συμφωνία και τώρα περιμένουμε να γίνει μια αλλαγή στην νομοθεσία και ότι θα επικυρωθεί ο καινούργιος νόμος τον επόμενο μήνα στη Σουηδία. Εδώ βλέπετε το προσωπικό μας. Δεν είναι βέβαια όλοι σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά σχεδόν. Πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε μια... δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις για 25 άτομα. Και τώρα μένουν 10 σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Μερικές φορές ε, προκυρήσουμε τις θέσεις. Οι πανδημίες μας απασχολούν πολύ. Νομίζω πάντως ότι προχωράμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας τώρα για την επόμενη χρονιά. Πρώτα απ' όλα έχετε πάρει αυτές τις πληροφορίες στους φακέλους σας, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στα σημαντικότερα σημεία. το σύστημα, οι οργάνους θα με απασχολήσουν στην παρουσίασή μου. Επίσης, επιδόσεις, δείκτες επιδόσεων για να βελτιωθεί το σύστημα, κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει των δραστηριοτήτων και επίσης εκατοχήρωση της ποιότητας και το σχετικό σύστημα. Αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία του οργανισμού μας και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με αυτά κατά προτεραιότητα. Ε, του χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες του. Ήδη μας έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Και με τα σας ανακοινώνω ότι ε, σε δύο εβδομάδες θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που μας έθεσαν. Τρία από αυτά τα ζητήματα είναι εγκάρσιου χαρακτήρα, το θέσω έτσι. Πρώτα απ' όλα, το θέμα των εργαστηρίων. Ε, με τη δημιουργία του οργανισμού μας ε, συζητήθηκαν τρία διαφορετικά πρότυπα. Ε, το πρώτο πρότυπο, το πρώτο μοντέλο ε, προέβλεπε πολλά εργαστήρια το δεύτερο, ένας μικρός οργανισμός ε, πρόληψης και ελέγχου νόσων ε, χωρίς εργαστήρια. Εγώ είχα ικανοποιηθεί με αυτό το μοντέλο γιατί ξέρω ότι υπάρχουν εξαιρετικά εργαστήρια στην Ευρώπη και δεν χρειάζεται επικάλυψη έχοντας νέα δηλαδή εργαστήρια στη Στοκχόλμη αλλά το, η αρνητική πλευρά είναι ότι ο οργανισμός μας ε, πρέπει να βασιστεί στα ε, υφιστάμενα εργαστήρια και αυτό με ανησυχεί. Γιατί ε, υπάρχουν περικοπές από πλευράς των εθνικών κυβερνήσεων ε, για τα εργαστήρια και αν συνεχίσουν οι περικοπές μπορεί τα εργαστήρια να μην είναι σε θέση να δίνουν αξιόπιστα δεδομένα στο ΕΚΠΕΝ, στο κέντρο μας. Οπότε του χρόνου θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με αυτά τα εργαστήρια για να συμφωνήσουμε σε ελάχιστες απαιτήσει που πρέπει να πληρούνται από τα εργαστήρια και θα δούμε πώς με αποτελεσματικό τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε τις απαιτήσει, τις εργαστηριακές απαιτήσει για την Ευρώπη και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Πιστεύω πώς είναι δυνατόν να εργαστούμε ε, πιο αποτελεσματικά. Ε, ένα από τα κοινά στοιχεία σε αυτά τα παραδείγματα που προέθεσα είναι ότι πλήττονται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από κάποιους νόσους, όπως η φυματίωση πλήττει τους φτωχότερους. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την υπατήτηδα, καθώς και τις νόσους που μπορούμε να προλάβουμε με εμβόλια. Πώς ε, λοιπόν αυτές τις περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες μπορούμε να τις προστατεύσουμε γιατί δυσανάλογα πλήττονται από τις μεταδοτικές νόσους. Ο πληθυσμός των Ρωμά. Ένα θέμα που σας απασχολεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι υποφέρουν από μεταδοτικές ασθένειες, από μολυσματικές νόσους. Θέλουμε του χρόνου να ε, δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις βέλτιστες πρακτικές, ε, ούτως ώστε να προστατεύσουμε αυτές τις πληθυσμιακές ε, ομάδες, πώς να αυξήσουμε το ποσοστό εμβολιασμών, παραδείγματος χάρη, σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα προλάβουμε πολλές νόσους ήδη από την παιδική ηλικία. Άλλο παράδειγμα, κλιματικές αλλαγές. Έχουμε αναπτύξει διάφορα σενάρια βάσει των οποίων ε, το κουνούπι τίγρης και η νόση που μεταδίδονται με τα τσιμπούρια θα φτάσουν και στην ίδια τη Στοκχόλμη. Με τις κλιματικές αλλαγές σαφέστατα θα επηρεαστεί η κατάσταση ως προς τις μολυσματικές νόσους. Λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους επαίοντε που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι σημαντικό. Οι εταίροι μας θα συμβάλλουν σημαντικά. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανάγκε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ποιε είναι οι δικέ σας ανάγκε, ποιε είναι οι ανάγκε των κρατών μελών και έτσι θα έχουμε τις σωστές κατευθυντήριε γραμμές για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Σας καλώ λοιπόν να τοποθετηθείτε κι εσείς και να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για αυτή την πρόσκλησή σας να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ε, η παρουσίασή σας και νομίζω ότι ε, θα ε, έχει γεννήσει πολλά ερωτηματικά στους συναδέλφους γιατί βλέπω ότι πληθαίνουν συνάδελφοι στα έδρανα. Η κυρία Γιανακουδάκη θα πάρει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. I forgot where the button was. Ε, που ήταν το σωστό κουμπί, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, ε, Dr. Springer, για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν. Ε, νομίζω έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ε, το περασμένο χρόνο. Έχουμε αρχίσει να ακολουθούμε τη σωστή ρότα. Βέβαια, υπολείπεται δύσκολο έργο, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Ερώτηση. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία ε, του κέντρου σας, ε, του ΕΚΠΕΝ. Ε, σε αυτό πρέπει να αποσκοπούμε. Γνωρίζω ότι έχετε συναντηθεί πολλές φορές με τους συντονιστές και έτσι έχετε διαμορφώσει μια άποψη σχετικά με τις ανάγκες του Κοινοβουλίου. Εδώ και πέντε χρόνια λειτουργεί το ΕΚΠΕΝ, αν δεν κάνω λάθος, πριν φτάσω εγώ στο Κοινοβούλιο και έχουν φύγει κάποια στελέχη ήδη Οπότε, ποιε μπορεί να είναι οι προσδοκίε, Νομίζω πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό τώρα. Για μένα αυτό συνιστά προτεραιότητα, εφόσον εσείς, ε, ε, εσείς είστε η επαφή μας. Τώρα, ε, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, στην Ελλάδα που θα μας ενημερώσει. Νομίζω θα πάω το Φεβρουάριο. Επίσης, επίσκεψη του Κοινοβουλίου και θα ήθελα ε, να ε, μεταβεί πολύ αριθμό κλιμάκιο εκεί για να καταλάβουμε πώς έχει η κατάσταση και τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την προσπάθεια. Χτες έγινε μία ακρόαση υπέρ των προβιωτικών. Δεν είναι ακριβώς μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΚΠΕΝ, αλλά είναι σημαντικό ε, γιατί ακούσαμε και την άλλη πλευρά, την άλλη επιχειρηματολογία, την αντίπαλη επιχειρηματολογία. Μα είπαν ότι το ΕΚΠΕΝ πρέπει να παρίσταται όταν έχουμε ακροάσει για να ακούνε ε, και την άλλη πλευρά και νομίζω ότι ήταν σημαντικές οι παρουσιάσει που ακούσαμε χτες. Λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε κάνει κάποιες καλές κινήσει, αλλά σίγουρα δεν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ε, σε ορισμένους τομεί. Μας μιλήσατε για τα εργαστήρια, μάλιστα. Πρέπει να δούμε και τι σχέσει με τα ε, λοιπά θεσμικά όργανα. Ε, για να εξοικονομήσουμε ε, χρόνο, χρήμα και να έχουμε και προστιθέμενη αξία. Πάντως, εν γέννη, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και περιμένω μια ανυπομονησία να ακούσω τις απόψεις και των συναδέλφων για να δούμε πώς θα ε, υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Πρόεδρος, η κυρία Ροτμπέρεντ έχει το λόγο. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. μετά από αυτά που ελέγχθησαν που καταδεικνύουν ε, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο για τον έλεγχο των ε, μολυσματικών ε, ασθενειών. Εμένα στο Κοινοβούλιο μ' αρέσει αυτό που ε, γίνεται που κατ' ε, είναι να ε, δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή να καταβάλλονται προσπάθειες που μερικές φορές είναι επώδυνες, αλλά εγώ θέλω να ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, επειδή εμείς εξετάζουμε σε βάθος το τι μπορούμε να κάνουμε με την αντιμικροβιακή αρρωγή. Μήπως ε, μπορείτε να δείτε, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Τι ακριβώς πιστεύετε ε, επ' αυτού. Βεβαίως και το θέμα της υγιεινής είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε μερικά νοσοκομεία η ταχύτητα της ε, νοσηλείας ε, και λόγω της έλλειψης προσωπικού ε, δεν υπάρχει διασφάλιση των απαραίτητων υγειονομικών συνθήκων. Μήπως ξέρετε και μπορείτε να κάνετε κάτι από αυτού όσον αφορά επίσης τα αντιβιωτικά. Πράγματι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον, αλλά δεν έχω και μια συγκεκριμένη λύση από αυτού. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για το 2011, μας προβάλλεται μια διαφάνεια, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς εννοείται με ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Thank you uh, very much. Um, Διάβασα τα πρακτικά παλαιότερων ε, συζητήσεων και κάποιος μίλησε για το περίφημο λογοπαίγνιο blame and shame. Κατά κάποιον τρόπο, δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί αυτό, αλλά δείχνει τις επιπτώσεις. Εμείς κατά κάποιον το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχει μια ασθένεια που μπορεί να προκληθεί από ένα ξενοδοχείο όπου, το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη του την ε, θερμοκρασία των υδάτων. Σήμερα το πρωί έγινε μια συζήτηση για τη διασυνοριακή υγεία. Η διασυνοριακή υγεία είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά μπορεί και να διευκολύνει την ε, διάδοση αυτών των ε, superbugs, των ιών που είναι ανθεκτικοί στα, μικροβι... αντιβιωτικά. Όταν λοιπόν ε, γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο και προσβληθεί κανείς από αυτόν τον ιό, μπορεί να μεταφέρει τον ιό αυτό σε άλλο νοσοκομείο, εφόσον χρειαστεί να επανεισαχθεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αυστηρές οδηγίες και να λαμβάνονται απαραίτητες πληροφορίες από τα νοσοκομεία. Μπορώ λοιπόν να σας δείξω στοιχεία για αντιμικροβιακή αντίσταση αναχώρα. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι εκείνο που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να αποκτήσετε πληροφορίες ε, με περισσότερες λεπτομέρειες και στην περίπτωση αυτή ε, θα μπορείτε να ελέγξετε ποια είναι η κατάσταση στις διάφορες ε, περιοχές και πάλι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί την αρχή συζητήσεων. Δεν είναι εύκολο αυτό. Νομίζω όμως ότι όλα ξεκινούν με το να δείξει κανείς τα γεγονότα και να δει ε, πώς μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Αυτό είναι το ένα. Και πρέπει να σας πω είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, όχι μόνο γιατί ε, απευθυνόμεθα στους ιατρούς αλλά και στους πολίτες να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όταν πάνε σε ένα γιατρό δεν χρειάζεται κάθε φορά να ζητάνε αντιβιωτικά γιατί μακροπρόθεσμα τα αντιβιωτικά δεν είναι δραστικά είναι λοιπόν είναι μια ε, προσέγγιση προς δύο ίσως και προς τρεις κατευθύνσεις και θα ήθελα στο μέλλον να συζητήσουμε το ποιες ε, θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες αυτής της ε, διασυνοριακής νέας πολιτικής και πώς μπορούν αυτή μπορεί αυτή η πολιτική ε, να επηρεάσει τις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Η τεχνογνωσία είναι το παν το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με το θέμα. Μιλάμε για ε, ιστούς, ε, κύτταρα του αίματος και όργανα και αυτά χρησιμοποιούνται για ε, μεταμοσχεύσεις και μπορούν να μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένα ε, τμήμα αυτών των ουσιών χρησιμοποιείται για τις ε, αποκαλούμενες ε, προχωρημένες θεραπείες. Υπάρχουν πάρα πολλές πολυκανονισμοί, νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χρήση τέτοιου είδους ιατρικών προϊόντων για προχωρημένες θεραπείες και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι αρμόδιος για αυτά τα φάρμακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ρώτησε πώς μπορεί να βοηθήσει στο να ελέγχεται καλύτερα η ε, μεταφορά των ασθενειών μέσα από ανθρώπινες ουσίες. Ξεκινήσαμε μία συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να δούμε πώς μπορούμε να εξετάσουμε από εκείνου τα θέματα. Έχουμε λοιπόν ε, ε, συντάξει ένα έγγραφο, ένα κοινό έγγραφο το οποίο στάλει στα διοικητικά συμβούλια των αρμόδιων οργανισμών και αυτό το έχω θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ποια είναι τα βήματα που προβλέπονται. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να εντοπιστούν οι απειλέ κατά την άποψή μας, να δούμε που ακριβώς μπορεί να ξεσπάσει μία νόσος. Δεύτερον, να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη και τους νέους φορείς. Και βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει είναι να χνηλατήσουμε τις ανθρώπινες ουσίες για να μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε την περαιτέρω διάδοση των ασθενειών. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον αυτό εντάσσεται ε, μέσα στην, ε, στις αρμοδιότητες που έχει το ΕΚΠΕΝ. Η απάντηση είναι μάλιστα διότι το ΕΚΠΕΝ καλύπτει τις απειλές στην ανθρώπινη υγεία από μολυσματικές ασθένειες και επίσης άγνωστης προέλευσης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα κάνουμε από κοινού με τον Οργανισμό Φαρμάκων. Γιατί ένα κομμάτι των ανθρώπινων ουσιών χρησιμοποιούνται ε, για φάρμακα. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά να τα κάνουμε μόνοι μας, πρέπει να τα κάνουμε σε συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ ε, που συμφωνήσετε κι εσείς ε, σε αυτό το κοινό έγγραφο. Από τεχνική σκοπιά, ο συνάδελφός μου, Τόμας Λάγκραντ και εγώ συμφωνήσαμε πάνω σε αυτή την πρόταση, αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι κατά πόσο θα συμφωνήσει από αυτής της πρότασης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για ένα ε, ιδιαίτερα περιεκτικό έγγραφο όπου μπορούμε να εξετάσουμε τα διάφορα θέματα και όπου μπορούμε να εξετάσουμε και τις αρμοδιότητες ε, που μπορούν να έχουν και οι διάφοροι φορείς, το ΕΚΠΕΝ και ε, ο Οργανισμός Φαρμάκων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σέρζιο Μπερλάτο έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ε, συγχαρώ τον δόκτωρα Σπρέγγερ και τον ε, και τους συνεργάτες του κέντρου για τη θαυμάσια εργασία που ε, προσφέρουν σε καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Στην έκθεση λοιπόν που είδα εγώ, εκεί δεν γίνεται καθόλου αναφορά και γι' αυτό θέλω να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις για το ενδεχόμενο μιας πανδημίας, κάτι το οποίο ευαισθητοποίησε πάρα σε τον τελευταίο καιρό. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην γρήπη των πτηνών και εν συνεχεία στην γρήπη των χείρων. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η Επιτροπή ανέλαβε μία σειρά πρωτοβολιών και θέσπισε μία σειρά μέτρων για να παρεμποδίσει τη διάδοση του ιού αυτών των ε, ε, ονομαζόμενων τότε πανδημιών που όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πανδημίες. Αυτές λοιπόν οι διατάξεις ε, εξακολουθούν να ισχύουν στην Ευρώπη και δυστυχώς περιορίζουν τις ε, οικονομικές ε, συναλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω ο κύριος Σπρέγκερ και το κέντρο του έχουν κάποια στοιχεία και ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά για να επικαιροποιηθεί η κατάσταση και για να κατανοήσουμε κατά πόσον έχει νόημα να διατηρούμε ακόμα τόσο αυστηρούς κανονισμούς οι οποίοι όπως σας είπα συνεχίζουν να επηρεάζουν πάρα πολλές οικονομικές συναλλαγές στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ροντμπέρεντ, έχετε μια ερώτηση. Έτσι δεν είναι. Παρακαλώ για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Σπρίγκερ μετά. Ναι. Ευχαριστώ. Έχω μιλήσει μαζί του έτσι κι αλλιώς και ιδιαίτερος, οπότε το ξέρει τι έχω να πω. Κοιτάξτε, επειδή τα είδαμε και σε διαφάνειες, θεωρώ ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για το 2011 για τις ουσίες αυτές, αλλά πρέπει να σας πω ότι εκπλήσωμαι για την ερώτηση της Επιτροπής. Από ό,τι έχω ακούσει εγώ από τον Γενικό Διευθυντή της Σάνκο. ήταν μια ιδέα. Εγώ βέβαια δεν έχω υπόψη μου κάτι γραπτό, πάντως πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την εντολή σας. Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνετε Το κοίταξα. Κοίταξα την εντολή σα για τι μεταδοτικέ ασθένειε και τα λοιπά. Σα το έχω πει πριν λίγε εβδομάδε. Υπογραμμίζω λοιπόν εδώ ότι θέλω να είσαστε προσεκτικό και να το κοιτάξετε αυτό το έγγραφο με πολύ προσοχή. Υπάρχουν ε, δεν είναι επειδή υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες που αλλάζουν και οι ευθύνες. Οι ευθύνε είναι έτσι όπως ε, τις ξέρουμε από τη δομή που έχουμε. Το λέω και προς τι γενικέ Διευθύνσει τη Επιτροπής. Πολύ προσοχή. Για το άλλο θέμα. Για την ιστορία αυτή του super bug, του υπερσκαθαριού και την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να το δείτε, γιατί αν όλο και περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτό, τι θα γίνει. Τι λέτε, ότι οι ασθενείς θα έρχονται στο νοσοκομείο και αν έχουν το μπαγκ αυτό θα μπαίνουν στην απομόνωση. Χρειάζεται να έχουμε και την κατάλληλη θεραπεία. Οπότε τι δυνατότητες υπάρχουν για θεραπεία, τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ιδέες έχετε και κίνητρα κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκασιεύσκα τώρα. E, Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά. Αυτά που είπατε από αυτά που είπατε, αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα είναι η απάντηση. Δηλαδή, που έλειπε, τι μέσα θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Είπατε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες περιπτώσεις υπατήτηδα ε, Β και Γ. Είπατε επίση ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε περιπτώσει φυματίωση, Είπατε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε περιπτώσει τροπικών ασθενειών. Όμω, δεν άκουσα τίποτα για την πρόληψη τέτοιων ασθενειών. Τι μέτρα πρόληψης λαμβάνεται για να ελέγχονται οι ασθένειες αυτές, γιατί ο οργανισμός σας ονομάζεται οργανισμός ο οποίος ελέγχει και προλαμβάνει νόσους. Οπότε πρέπει να πούμε εδώ ότι οι γονείς νεογέννητων προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των εμβολίων τα οποία κάνουν τα παιδιά τους. Αυτό απορρέει από μια αρνητική εκστρατεία που λέει ότι ο εμβολιασμός μπορεί να μειώνει την αντίσταση των παιδιών, μπορεί να δημιουργεί κάποιες ασθένειες κλπ. Εσείς το έχετε δει καθόλου αυτό το πρόβλημα, το έχετε εξετάσει. Ο οργανισμός σας σκοπεύει να κάνει μια εκστρατεία στους γονείς έτσι ώστε οι γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους γιατί το εμβολιασμό προλαμβάνει τις ασθένειε. δεν τις προκολεί. Η κυρία Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξή. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που καθυστέρησα, μπορεί να το είπατε και να μην το άκουσα εγώ. Πάντως, για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες και τις τοπικές ασθένειες. Υπάρχουν υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Εφόσον συνεργάζονται, και ελπίζω ότι συνεργάζονται, τότε μπορούμε να έχουμε τέτοια στοιχεία. Όμως συχνά αντιμετωπίζω προβλήματα. Συχνά τέτοιες πληροφορίες δεν ζητάτε μόνο εσείς, αλλά ζητάει και ο ΠΟΗ, ζητάνε και άλλοι οργανισμοί είναι ερωτηματολόγια ιδιαίτερα μεγάλα, πληρέστατα και πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη στην ενημέρωση. Τα διάφορα λοιπόν κέντρα και αισθητούτα των κρατών μελών δυσκολεύονται να καλύψουν ε, τη ζήτηση. Αν λοιπόν υπάρχει όντω επικάλυψη, δεν θα μπορούσατε να φροντίσετε να συνεργάζεστε καλύτερα με άλλους παγκόσμιους οργανισμούς για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας αλλά και το οικονομικό κόστος που επιφορτίζονται οι εθνικοί αυτοί οργανισμοί. Μπορείτε να μας πείτε αν σχεδιάσετε κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο. Πέρα από αυτά που εσείς ζητάτε αλλά και άλλοι οργανισμοί, μερικές φορές λείπει η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος ε, Λούκας Αρτόγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τις ασθένειες, την φυματίωση για παράδειγμα. Ε, Πώς λαμβάνετε εσείς υπόψη σας την επικουρικότητα, ο οργανισμός σας δηλαδή, γιατί πολλές φορές τα κράτη-μέλη έχουν αντίστοιχου οργανισμού. Τι γίνεται με την επικουρικότητα. Έπειτα, εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Προπολογισμών και έχουμε διαπιστώσει στις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση του οργανισμού σας. Ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Και αναρωτιέμαι μήπως ο οργανισμός σας έχει κάποια σχέδια για να βελτιώσει το θέμα της οικονομικής διαφάνειας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χάρτογκ. Ο τελευταίος ελέγχθησαν ε, αρκετά από αυτά που θέλω να πω, κυρίως από τον συνάδελφο Μπερλάτο, που ζήτησε κάποιες ε, διευκρινήσεις ε, και είπε γιατί δεν αναφέρονται τα στοιχεία για τις ε, υποτιθέμενες πανδημίες ε, που τελικά απεδείχθησαν απλά ε, κάποιες επιδημίες. Δεν πρέπει λοιπόν να τα πανάμε άσκοπα τα κονδύλια και να ανησυχούμε τους πολίτες, όπως ακριβώς απεδείχθη σε αυτούς τους ε, δύο, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που ήταν φήμες παντελώς αβάσιμες. Όσον αφορά τώρα την ε, παγκοσμιοποίηση, ξέρουμε ότι η μετακίνηση ατόμων και εμπορευμάτων από τρίτες χώρες συνεπάγεται όχι μόνο τη μεταφορά ιών και ασθενειών, ε, κυρίως της ελονοσίας ή της φυματίωσης μάλλον, της φυματίωσης, αλλά ε, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ζώα που μεταφέρουν σε κοντένερ και που μπορούν αυτά να μεταφέρουν ασθένειες. Υπάρχουν ενέδρε τσιμπουριών, υπάρχουν ε, οι μύγες, τα κουνούπια και το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να συμπεριφερθεί για να περιοριστεί ο κίνδυνος οι Ευρωπαίοι πολίτες να ε, πληγούν από αυτές τις μολυσματικές ασθένειες που κάποτε ήταν άγνωστες στην Ευρώπη. Τι προτίθεστε λοιπόν να κάνετε και για το θέμα του εμβολιασμού. Γιατί πάρα πολλές ασθένειες ξεκινώντας από την ε, υπατήτηδα, εν πάση υπάρχουν ε, ε, πολλές ασθένειες που είναι σημαντικές όπως η μηνυγκίτης, παραδείγματος χάρη, μπορούν σήμερα να προληφθούν με εμβολιασμό. Εμβολιασμός που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη, άμα στην, στην Ιταλία όμως ε, κάποια ε, εμβόλια είναι δωρεάν, αλλά πάλι όχι. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σημαντικές συνέπειες, ε, διότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε δωρεάν εμβολιασμό ή έστω να ενημερωθούν ότι οι εμβολιαζόμενοι αποφεύγουν κάποιες ασθένειες που μπορούν να αποβούν και μοιραίες. Και κλείνω με το εξή αίτημα. Εσείς έχετε αξιολογήσει ε, τη δυνατότητα να ζητήσετε και επιμένω να ζητήσετε γιατί τελικά η τελική αρμοδιότητα εναπόκειται στα κράτη-μέλη ε, να ασχοληθείτε με το σύνδρομο το ε, πολλαπλό χημικό. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο συνεπάγεται πάρα πολλά προβλήματα σε όσους πληγούν από αυτό το σύνδρομο. Είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι γίνεται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάντως όποιο πλήττεται από αυτό το σύνδρομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πλέον τίποτα που να περιλαμβάνει χημικέ ουσίε. Και αυτό συνεπάγεται τεράστια προβλήματα για τη διατροφή του ανθρώπου αλλά και για τη ζωή του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το κινητό τηλέφωνο, ούτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν μπορεί να ζήσει καν σαν φυσιολογικό άνθρωπο. Και στην ιταλια δυστυχω δυστυχώς μόνο δύο-τρει περιοχέ αναγνωρίζουν αυτή την ασθένεια ω αναγνωρισμένη ασθένεια και δίνουν τα φάρμακα δωρεάν. Και στην περίπτωση αυτή ερωτώ, ε, προτίθεστε να παρακολουθήσετε και αυτήν την ασθένεια όπως και άλλες ασθένειες που είναι σπάνιες αλλά αυτή δεν γίνεται πια τόσο σπάνια για να υπάρξει κάποια παρέμβαση κυρίως υπέρ εκείνων των ανθρώπων που υποφέρουν όχι διότι έχουν πληγεί από μια ασθένεια που είναι λιγότερο ε, αξιοσέβαστη από άλλες, αλλά διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες θεραπείας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια στοιχεία πριν ζητήσω από τον κύριο Σίγκερ να μας απαντήσει. Τον κύριο Σπρέγκερ ζητώ, συγγνώμη. Οι συνάδελφοι μίλησαν για τη γρήπη ή τα νιένα. Ε, εκπονείται τώρα μία εκθεσή και εμείς έχουμε εδώ διοργανώσει στο Κοινοβούλιο διάφορες ακροάσεις. Χτες εξάλλου η κυρία Ριβεζιέ και οι ε, διοργανώσαμε μια σχετική ακρόαση, άλλη προβλέπεται για το Δεκέμβριο. Λοιπόν, θέλουμε να ερωτήσουμε το εξής τον κύριο Σπρέγκερ. Για ποιο λόγο, ε, παρά την αξιολόγηση που είχε κάνει το ΕΚΠΕΝ για την πανδημία, ε, της η οποία ήταν και ιδιαίτερα λογική και ε, η οποία δεν συνέστη ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή δεν ανέφερε ότι υπήρχε σοβαρός λόγος ανησυχίας. Γιατί λοιπόν με φρενήρις ρυθμούς αγοράστηκαν τα εμβόλια που τελικά χρησιμοποιήθηκαν από υγιείς ενήλικες πριν από ένα χρόνο ε, στην ίδια αίθουσα αυτά συζητούσαμε. Λοιπόν, έγινε αυτή η μετροπαθής αξιολόγηση. Αλλά τελικά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ακολούθησαν αυτή την αξιολόγηση ανταυτής. Βασίστηκαν στην πολύ πιο απεσιόδοξη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και γνωρίζουμε όλοι ε, τις ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, αυτής της απόφασης. Thank you very much for Πάρα πολλές ερωτήσεις. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για αυτό το ζήτημα. Πρώτη ερώτηση. για το σχέδιο δράσης για την πανδημία. Τι είναι το πιο σημαντικό. Να γίνει σωστή αποτίμηση του κινδύνου. Να μην υπερβάλλουμε ως προς τον κίνδυνο, διότι ενδέχεται αυτό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο. Θα πρέπει να βασιστούμε στα πραγματικά στοιχεία. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Οι αξιολόγησεις κινδύνου ε, είναι ε, ισόρροπες, αυτές που δημοσιεύει δηλαδή το κέντρο μας. για τις ε, ουσίες, τις ανθρωπογενείς ουσίες, ανθρώπινης προέλευσης, SHO. Η κυρία Ροτ έθεσε ένα σχετικό ερώτημα και μάλιστα Μα ρωτήσατε συγκεκριμένα γιατί δεν ε, συνεργαστήκαμε περισσότερο με τον ΕΟΦ. Ε, μα είχε υποβληθεί το αίτημα να εκπονήσουμε εμεί ένα σύστημα από πλευρά ΕΚΠΕΝ. Είχαμε συμφωνήσει για μια κοινή προσέγγιση, είχαμε κάνει και υπολογισμό του κόστους και μπορέσαμε να ε, τον ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα εργασιών μας, ε, στο σχέδιο δράσης. Αλλά ποια είναι η απάντηση που πήραμε. Αποκλείεται. Χρειαζόμαστε νέο προσωπικό, χρειαζόμαστε νέα κονδύλια. Εφόσον όμως ε, γίνονται περικοπές στους προϋπολογισμούς, δεν μπορούμε εμείς να ζητούμε επιπρόσθετα κονδύλια Ενσωματώσαμε το επιπρόσθετο κόστος λοιπόν στο πρόγραμμά μας και τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών μας. Ε, μπορώ να σας κοινοποιήσω και το έγγραφο που υποβάλαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι το έγγραφο εργασίας μας. Για το Superbug, αυτό το πολύ ανθεκτικό ε, ιό ε, του Νέου Δελχή συγκεκριμένα, έχουμε κάνει αποτίμηση κινδύνου και είναι σαφές ε, ότι η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Συζητήσαμε με πολλούς εμπειρογνώμους από εργαστήρια πώς μπορούμε να επιτύχουμε έγκαιρη, ε, ταχύτερη διάγνωση. Ε, συμφωνήσαμε επί κάποιων μεθοδολογιών και την πραγματογνωμοσύνη την μοιραστήκαμε με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι γιατροί έχουν επίγνωση των προβλημάτων κυρίως αν ο ασθενής ε, έχει πάει στην Ινδία. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, να τους ευαισθητοποιήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Ποια, ποιο είναι το αποτέλεσμα τώρα. Αν μολυνθείτε από αυτό το πολυανθεκτικό μικρόβιο, μόνο δύο αντιβιωτικά ε, είναι αποτελεσματικά είναι αποτελεσματικά, αλλά έχουν ισχυρότατες παρενέργειες και παρουσιάζουν και άλλες δυσκολίες. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερω που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ε, προωθεί ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα για νέα αντιβιωτικά. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή από πλευρά τη Επιτροπής επαναλαμβάνω ότι το ΕΚΠΕΝ δεν ε, ε, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του κινδύνου. Εμεί κάνουμε αποτίμηση κινδύνου. Δίνουμε τα τεκμηρία, τα στοιχεία και κατόπιν τα κράτη-μέλη, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν τις αποφάσεις. Ε, υπάρχει αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων ε, που με ικανοποιεί εμένα γιατί αν ε, ληφθεί απόφαση για εμβολιασμό και πρέπει να αποφασιστεί το σχετικό κονδύλιο δεν μπορεί το ΕΚΠΕΝ χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κονδύλιο να αποφασίσει για τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού είναι πολύ καλό που υπάρχει κατανομή των αρμοδιοτήτων όσο έχει τώρα. Δεν έχουμε δηλαδή τα απαιτούμενα μέσα για να επιβάλλουμε μέτρα και μετρήσεις σε διάφορες χώρες. Ε, για τους εμβολιασμούς των παιδιών έχουμε όντως ε, προγράμματα για να αυξήσουμε την ε, ενημέρωση και να μελετήσουμε ε, ποιο είδους πληροφορίες είναι ε, πλέον αποτελεσματικές. Για τη γρήπη έχουμε μάθει πολλά πράγματα, γιατί ε, το ένα από τα προβλήματα είναι η ελλειπής ενημέρωση. Αν θέλετε λοιπόν να προστατεύσετε όχι μόνο τους πλουσίους, αλλά όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, χρειάζεστε καλές πληροφορίες. Και οι καλές πληροφορίες δεν διανύμονται με επιστολές. θυμάστε το, ε, HPN, χρειαζόμαστε και τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον. Αναφερθήκατε στον ε, ΠΟΗ. Ε, πολλά ερωτηματολόγια εστάλησαν ε, στα κράτη-μέλη και από το ΕΚΠΕΝ είναι σημαντικό να δούμε πώ θα επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό. Διότι αυτό συνεπάγεται ε, δυσανάλογα μεγάλο άχθο για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή να ε, αποστέλουν απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτηματολόγια. Νιώθω κι εγώ υπεύθυνο. Ε, συνεργαζόμαστε στενά ε, με τον ΠΟΗ, τον Παγκοσμίο Οργανισμό Υγεία, ε, για όλα αυτά τα ζητήματα. και θα μελετήσουμε πώς μπορούμε να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας χωρίς επικαλύψεις. Τα, οικονομικά, το, τα ερωτήματα οικονομικής φύσης. Ε, μπορώ να σας δώσω με τα χαράς οικονομικά στοιχεία, γραπτός κιόλα. Μπορείτε να σας κοινοποιήσω τον προϋπολογισμό, όλα τα επιμέρους ε, τμήματα και κεφάλαιά του. Μας ε, ρωτήσατε για την προσθέμενη αξία του ε, ΕΚΠΕΝ. Πριν από έξι χρόνια μας ρωτήσατε γιατί χρειαζόμαστε το ΕΚΠΕΝ. Τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε ο ιός SARS. Και ήταν σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών. Αυτό κάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, παρότι είναι μικρό, είναι μια μικρή οντότητα, ε, προσπαθεί να ε, επιτύχει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε επίπεδο κρατών μελών και ε, αποφεύγοντας έτσι τις επικαλύψεις. Για την γρήπη το αποδείξαμε ότι προσφέρουμε προς τη θέμενη αξία. Πάντοτε σας ενημερώναμε για την κατάσταση είναι ιδιαίτερα οι ισόρροπες που έδινε η προηγούμενη διευθύντρια και ποτέ δεν υπερέβαλε σε σχέση με τις προσδοκίες, δηλαδή για τις ενδυνάμει επιπτώσεις ε, της ε, γρήπης. Ένα άλλο ερώτημα είχε σχέση με το κτίριο. Το νίκη για το κτίριο, τη μίσθωση του κτίριου. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει απευθύνει ιδιαίτερε επικρίσει ε, για το νέο μας εκτίριο και είχα χαρεί και εγώ ε, τρόπον την με αυτή τη δήλωση διότι έτσι ξεκίνησε η συζήτηση ε, και συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις σας. Εξάλλου τώρα ε, αναζητούμε ένα ε, δικτύριο ε, χαμηλότερου κόστους και εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια. Ε, προφανώς υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου, υπάρχει και εσωτερική υπηρεσία ελέγχου, υπάρχει και το ελεγκτικό συνέδριο. Όλοι ελέγχουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού μας και δεν θα εμποδίσουμε κανέναν. Όλοι ευπρόσδεκτοι. για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων. Ε, υπάρχει ο Διεθνής Κανονισμός Υγιεινής ε, που γίνεται σεβαστός. Ε, συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τους κτηνιάτρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλές εμολυσματικές νόσοι είναι ζωνόσοι, δηλαδή προκαλούνται από τα ζώα και είναι αγαστή η συνεργασία μας με τον κτηνιατρικό τομέα. Άλλη ερώτηση για τις διαφορετικές πολιτικές εμβολιασμού, συγκεκριμένα για τα παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το ερώτημα. Πώς να το θέσω. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για τα προγράμματα εμβολιασμού. Εσείς μιλήσατε για διασυνοριακή υγεία. Όταν Διασχίζεται τα σύνορα, ισχύει διαφορετικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Ε, αυτό προξενεί κατάπληξη. Αλλά ποια είναι τα επιστημονικά τεκμήρια. Καλό θα ήταν να γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, για το ΝΙΤΑ 1 1 την πανδημία. Πολύ δύσκολη ήταν η ερώτησή σας, ε, Πρόεδρε. Εμείς δώσαμε τα στοιχεία, την ε, αξιολόγηση κινδύνου και οι πολιτικοί ηθήνοντες, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, πρέπει να ε, επομιστούν τι τους για τη διαχείριση του κινδύνου. Εγώ δεν δύναμε να το σχολιάσω το ζήτημα. Αναμένουμε τα πορίσματα του εργαστηρίου της κυρίας Δρυβαζή ήταν πολύ χρήσιμο που διοργανώθηκε, χρειαζόμαστε πληροφορίες και ελπίζουμε να αντλήσουμε διδάγματα. Ε, κατά τη διάρκεια της ακροάσεως, εγώ προσωπικά άντλησα τρία διδάγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε καλύτερη αποτίμηση κινδύνου. Υπάρχει νέος ιός όταν υπάρχει νέος ιός συγγνώμη, και πώς μπορούμε να προβλέψουμε τις συνέπειες για να έχουμε καλύτερη διαχείριση κινδύνου μετά την αξιολόγηση κινδύνου και ε, να έχουν και οι ε, πολιτικοί φορείς ε, καλύτερα στοιχεία στη διάθεσή τους για να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τη διαχείριση του κινδύνου και πρέπει να συνυπολογίσουμε διάφορους παράγοντες κοινωνικούς, οικονομικούς και αλλού όχι μόνο τα βιολογικά δεδομένα. Τώρα, η επικοινωνιακή πολιτική πώς με αξιόπιστο τρόπο θα επικοινωνούμε με τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνιστά μεγάλη πρόκληση προς το παρόν. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροτμπέρεντ, νομίζω ότι έχετε κάτι να πείτε. Ναι. Δεν ξέρω κύριε Σπρίνγκ αν είναι έτσι, αλλά οι δημόσιες ε, συνεδριάσεις δεν είναι τόσο καρποφόρες όπως οι κατηδίαν που έχουμε. Θα επανέλθω σε κάτι. Φυσικά και ξέρω ότι εσείς διαχειρίζεστε, ήμουν εδώ πέρα και όταν ετοιμάσαμε το καταστατικό της, ε, του οργανισμού σας. Αλλά υπάρχει μια διαφορά με το εμάς, διότι κάνουν, ε, προετοιμάζουν και τις άδειες για τα φάρμακα. Αυτή είναι η διαφορά με το δικό σας τον οργανισμό. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο απτά στη δικιά σας περίπτωση. Και ίσως, όπως και ο συνάδελφος από την Ολλανδία, να νομίζουν ότι είναι περιττός ο σας. Δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ότι αυτό οφείλεται επειδή υπάρχει ο ΠΟΗ. Ο ΠΟΗ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες που υπάρχουν για να δούμε τι συμβαίνει σε ολόκληρο το κόσμο. Πιστεύω ότι έχετε διαφορετικό ρόλο. Οι άλλες ε, αρχές έχουμε εμείς, άλλες εισήνουν για την Αφρική. Πάντως, για να επανέλθω στο τι μπορούμε να κάνουμε για το περίφημο Super Bug. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, πείτε μου τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει ερευνητικά προγράμματα. Εγώ το ξέρω, αλλά γιατί δεν μας το λέτε. Δεν χρειάζεται να μας στείλετε τίποτα, εγώ το έχω. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτιάχνει φάρμακα, εντάξει η έρευνα, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε και πιο πέρα και να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Και για να επανέλθω και στο άλλο, Εξακολουθώ να πιστεύω, όσον αφορά την εντολή σας, ότι τίποτα δεν υπάρχει στην εντολή σας που να σας επιτρέπει να ασχολείστε με ουσίες ανθρώπινης ε, προέλευσης. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να το δούμε διαφορετικά αυτό. Θα το ξανακοιτάξω πάντως το κείμενο. Θα το δω και με τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο για να φροντίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει λόγο όταν έχουμε να κάνουμε με τον ρόλο του οργανισμού σας, του ΕΚΠΕΝ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Θέλω να απαντήσω. Γιατί το να μιλάμε για το EMA και για τα φάρμακα, για την υπηρεσία για τα φάρμακα δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτού. Το ερώτημα είναι ποια είναι η εντολή όταν έχουμε να κάνουμε με τη δημόσια υγεία. Και βεβαίω και θέλω και εγώ να συνεισφέρω στη συζήτηση για την μελλοντική μας εντολή. Και θα γίνει. Διότι θα γίνει συζήτηση για την εντολή μας και ελπίζω, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ανοιχτή σε παντό είδου επιχειρήματα. Πάντως θα ήθελα να συζητήσω και μαζί σας και με την ομάδα για την υγεία ποιο θα είναι το μέλλον της εντολής της υγείας. Όσον αφορά τώρα τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, δύο παραδείγματα έχω τον ε, πυρετό Q στην Ολλανδία, όπου εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα όταν συζητούσαμε για τις μεταγγίσεις αίματος. Όταν υπάρχει τέτοιος πυρετός, ε, μπορούμε να κάνουμε μεταγγίσεις. Και για άλλους ιούς επίσης έχει τεθεί ε, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν ότι ταιριάζουν με την εντολή μας. Είμαι όμως ανοιχτός προς συζήτηση. Και υπάρχει και πολιτική συζήτηση βέβαια για το τι προσέγγιση θέλετε να ακολουθήσετε όσον αφορά τις ουσίες αυτές. Τώρα από τη δικιά μου την πλευρά μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε φτιάξει αυτό το έγγραφο εργασίας και είμαι πεπισμένος ότι είναι αξιόπιστο. Αυτή είναι η δικιά μου ευθύνη. Από εκεί και πέρα το πολιτικό επίπεδο θα αποφασίσει κατά πόσο το θέλει ή δεν το θέλει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Μπερλάτο, έχετε ζητήσει να κάνετε μια ερώτηση ακόμα. Πρόεδρε, θα ήθελα να επέμβω για άλλη μια φορά, γιατί Προηγουμένως ευχαρίστησα τον Δόκτωρα Σπρέγκερ και το κέντρο για τη δουλειά που κάνουν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος με την απάντηση που μου δώσατε. Έκανα μια ερώτηση και δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Σπρέγκερ δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να απαντήσει. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να την επαναθέσω, ίσως να είναι πιο κατανοητή τώρα. Η γρήπη των πτηνών αφορά έναν ιό που είναι γνωστός ε, εδώ και αρκετό καιρό στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη γρήπη των ε, πτηνών θα αναγκαστούμε να ζούμε τους επόμενους αιώνες και επειδή αυτή η γρήπη τελικά δεν αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Δεν αναφέρομαι στην υγεία των πτηνών. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι όλα τα μέτρα που ελήφθησαν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που προέκυψαν ως ε, υπερβολικά μέτρα Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα οποία διαπιστώσαμε και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι υπάρχουν ακόμα μέτρα και προφύλαξη που ισχύει και επιβαρύνουν κατά πολύ τις δραστηριότητες και όχι μόνο οικονομικές. Ερωτώ λοιπόν, μήπως μπορείτε εσείς να προβείτε σε μια αξιολόγηση για αυτά τα οποία συνέβησαν έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε στους πολιτικούς χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να ε, διαπιστώσουν και εκείνοι ότι ορισμένα μέτρα τα οποία ισχύουν ακόμα είτε να χαλαρώσουν είτε να καταργηθούν πλήρως. Μήπως ε, μπορείτε να μου αναφέρετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί έχω τελείψει ότι κάτι πενήσεστε και προσπαθώ να ε, καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε, αναφέρομαι παραδείγματο χάρη στο εμπόριο ε, ζώων ή ε, της, των πτηνών, του δέρματος των πτηνών των φτερών των πτηνών αναφέρομαι ε, στην ε, απαγόρευση κυνηγιού εκτός ε, από ορισμένε εξαιρέσεις. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια στοιχεία που εξακολουθούν να ισχύουν και δεν είναι τεκμηριωμένα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και ότι δεν προέκυψε τελικά πανδημία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα νέο ιό όπως αυτός στον οποίο αναφέρθηκε ο προλαλής σα. Γνωρίζουμε εδώ και αιώνε τον ιό αυτό, γνωρίζουμε την επικινδυνότητά του για τα ζώα και όχι για για τους ανθρώπους δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστεί με υπερβολικό τρόπο μια υποτιθέμενη πανδημία η οποία όπως το έχουμε προβλέψει τελικά δεν προέκυψε μήπως λοιπόν μπορούμε να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα όσον αφορά το θέμα αυτό ή θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο το επίπεδο συναγερμού Κατανοώ την ε, ερώτησή σας. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να έχω περισσότερες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας δώσω μια αξιόπιστη απάντηση και δεν την έχω πρόχειρη. Πρέπει λοιπόν να μιλήσω στους συνεργάτες μου για να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας Oui. Άλλες ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Χανόγκ. Θα ήθελα να είναι διαθέσιμα γραπτά τα στοιχεία, τα οικονομικά του ΕΚΠΕΝ για να είναι σίγουρη η νομιμότητά του. Θέλουμε να υπάρχει εγγύηση ότι έχουμε τα στοιχεία. Πρέπει να μπορούμε να τα δούμε και να αξιολογούμε σε συνεχή βάση κατά πόσο είναι εντάξει. Να μας τα στείλετε λοιπόν. Παρακαλώ για να τελειώσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο στον ε, κανονισμό. Αναφέρεται ότι κάθε πέντε χρόνια θα υπάρχει μια εξωτερική αξιολόγηση και η επόμενη θα είναι το 2012. Δεν είναι μόνο το SARS, ε, πρέπει να πάμε και 50 χρόνια πίσω. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε περίπου 20 δίκτυα για συγκεκριμένες ασθένειες. Αυτό λοιπόν κόστισε πάρα πολλά χρήματα και ένας από τους λόγους ήταν για να υπάρξει εναρμόνιση, ε, να γίνει εξοικονόμηση κονδύλιων και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομήσαμε αρκετά κονδύλια και έχουμε αρκετές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που σας έδειξα για ασθένειες σε διάφορες χώρες, αυτές οι πληροφορίες δεν υπήρχαν μέχρι πριν από τρία χρόνια. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ορισμένες χώρες πρέπει να εργαστούν σκληρά για να ελέγξουν τις μολυσματικές ασθένειες. Και το θέμα είναι ότι οι ασθένειες αυτές ε, μπορεί να είναι και διασυνοριακές. Δηλαδή αν δεν προσέξει ο γείτονά σα, ε, θα υποφέρετε και εσείς από την ασθένεια αυτή. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με ε, χώρες που θα μπορούσαν να πληγούν με τις υποψήφιες χώρες, με με τις υποψήφιες χώρες για να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις μολυσματικές ασθένειες. Πάντως μπορείτε κάλλιστα να έρθετε να μας επισκεφτείτε και φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να σας πείσω σε μια επιτόπια επίσκεψη. Δόκτωρα Σπρέγγερ, εκ μέρου τη Επιτροπή μα ολόκληρη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, που ήταν καρποφόρα, χωρί ξύλινη γλώσσα. Ίσως γιατί δεν ήμασταν φοβερά πολύ άριθμοι. Μπορέσαμε λοιπόν να υποβάλουμε πολλέ ερωτήσει, πήραμε και πολλέ απαντήσει. Οπότε, εκ μέρου όλων των συναδέλφων, σα ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Τα σημεία 9 και 10 θα εξετάσουμε τώρα και μετά το σημείο 8. Αλλά λίγα λεπτά διακοπή για να συνοδεύσω στην έξοδο των ε, προσκεκλημένων μας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 9 της ημερήσια διάταξη, που είναι η επικύρωση και νομική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τι δοκιμέ σε ζώα στον τομέα των καλλιντικών. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος εσεί, η κυρία Λεκρενιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ για να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε την έκθεσή μας όσον αφορά τις εναλλακτικέ μεθόδους που μπορούν να υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα στο τομέα των καλλιτικών. Και αυτό για την περίοδο 2007 και 2008 είναι η 8η έκθεση που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα μιλάει για την, ε, τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βεβαιωθούμε ότι είναι αυλαβή τα καλλικαντικά. Επίσης αναφέρεται εκεί και τα ίδια των πειραμάτων που ακολουθούμε. Έπειτα υπάρχουν οι εναλλακτικέ μέθοδοι που μπορούν να υποκαταστήσουν ε, πειράματα στα ζώα και που ισχύουν σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Την έκθεση αυτή την ετοιμάσαμε βάσει του άρθρου 9 τη οδηγία για τα Καλλιντικά. Έχει την εξή ιδιαιτερότητα είναι η τελευταία που καλύπτει την περίοδο πριν από την 10η Μαρτίου 2009, γιατί τότε άρχισαν να ισχύουν η πλήρης να ισχυουν οι πληρης απαγορευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πειραμάτων σε ζώα για καλλιντικά, καθώς επίσης και απαγόρευση εμπορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιντικών που έχουν χρησιμοποιήσει σαν πειράματα ή τα συστατικά τους έχουν πειραματιστεί σε ζώα. Εκτός όταν πρόκειται για την τοξικότητα, την επανειλημμένη τοξικότητα των προϊόντων αυτών. Θα σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για το περιεχόμενο της έκθεσης και μετά θα έρθω στις σημερινές μας δραστηριότητες τις σχετικές με τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής. Το πρώτο τμήμα τη έκθεσης αναφέρεται λοιπόν στα πειράματα που γίνονται στα ζώα. 27 χώρες μέλη έχουν δώσει πληροφορίες από αυτού. Βάσει των στοιχείων αυτών, καλλιντικά έχουν χρησιμοποιήσει πειράματα σε ζώα και το 2007 και το 2008 στη Γαλλία και στην Ισπανία. 1500 για το 2008 και από τότε που έχουμε τα στατιστικά δεδομένα έχουμε διαπιστώνει ότι το 2004 είχαμε 6.000 ζώα, ήταν χρονιά που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο πειραματόζωα. Για να διευκολυνθεί τώρα ο υπολογισμό και για να έχουμε τέτοια στοιχεία, η Επιτροπή έστειλε κατευθυντήριε γραμμέ στα κράτη-μέλη. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτησε τα κράτη-μέλη για τι μεθόδου που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ελέγξουν την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων, τέτοιων προϊόντων, όπως προβλέπεται από τις 11 Μαρτίου, όπως είπαμε, του 2009. Και προτείνονται επίσης και αναλλακτικέ μέθοδοι. Η έκθεση αναφέρει μεθόδους που νομικά είναι αναγνωρισμένες και αναφέρει επίσης και τις επιστημονικές πρόοδους που έχουν επιτευχθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων, αναγνωρισμένων εναλλακτικών μεθόδων. Έτσι λοιπόν από το 2009 υπάρχουν ε, άλλες μέθοδοι που υποκαταστούν τις δοκιμές σε ζώα, εκτός όπως είπαμε για την περίπτωση της τοξικότητας. Έχουν αναγνωριστεί λοιπόν από την οργάνωση αυτή πολλές ε, τέτοιες μέθοδοι, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε υποκαταστήσει πλήρως τα πειράματα ε, στα ζώα. Τα πειράματα για τα οποία από το 2013 τώρα θα απαγορευτεί η εμπορία προϊόντων που έχουν χρησιμοποιήσει δηλαδή τέτοια πειράματα, εδώ η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Η έκθεση αναφέρεται στα συμπεράσματα της εκφάμου. Εναλλακτικές λύσεις δεν έχουμε, όμως υπάρχει πρόοδος και γίνονται ακόμα ερευνητικέ προσπάθειες που στηρίζονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κόλυπα με 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε διεθνές επίπεδο η συνεργασία για τις αναλλακτικές μεθόδους έχει προχωρήσει πολύ έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο για την συνεργασία σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις μεθόδους που υποκαταστούν πειράματα με ζώα. Η συμφωνία αυτή έγινε το Σεπτέμβριο του 2008 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Είναι συμφωνία που ευνοεί την συνεργασία σε θέματα επιστημονικής έγκρισης εναλλακτικών μεθόδων. Μετά την περιγραφή αυτή του περιεχόμενου της έκθεσης θέλω να πω δύο λόγια και για το τι κάνουμε σήμερα προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή τα συμπεράσματα της έκθεσης. Στην επόμενη έκθεση θα επικεντρωθούμε στο θέμα της εφαρμογής των απαγορεύσεων. Όπως επίσης θα δούμε και τι εναλλακτικέ μέθοδοι υπάρχουν. Το κύριο σημείο θα είναι τα πειράματα που περιέχονται στην απαγόρευση που θα αρχίσει να ισχύει από το 2013. Η οδηγία αναφέρει την τοξικότητα σε επανελμένες δόσεις και την αναπαραγωγική τοξικότητα. Θα ήθελα εδώ να σταθώ λίγο στην επιστολή που έστειλε η Επιτροπή σας στο κοινικό μας διευθυντή πρόσφατα. Ε, ζητούσατε να σας ε, πούμε ποιος είναι ο ορισμός των ενιών αυτών. Πάμε λίγο πίσω, το 2003. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να ετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα βάσει της οδηγίας για την εφαρμογή της απαγόρευσης εμπορίας. Η Επιτροπή έτσι ετοίμασε μια ομάδα ad hoc με μερικούς επιστημονικούς εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, τις οργανώσεις που προστατεύουν τα ζώα και τις κυβερνήσεις. Η ομάδα αυτή εκπώνησε έκθεση καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για την εξαφάνιση των πειραμάτων ε, με ζώα για τη δημιουργία καλλιντικών. Στη συνέχεια το 2009, τον Ιούλιο, η ομάδα αυτή ενέκρινε μία γνωμοδότηση. Και βάσει της νομοδότησης και της έκθεσης, οι υπηρεσίε της Επιτροπής δημοσίευσαν ένα έγγραφο εργασίας που φέρει ως τίτλο «Χρονοδιάγραμμα για το phasing out των πειραμάτων με ζώα βάσει της 7ης τροπολογίας της οδηγίας για τα καλλιντικά». Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται διάφορα σημεία ανάλογα με τις προθεσμίες που αντιστοιχούν σε αυτά. Το endpoint, η τοξικότητα επανειλημμένα καλύπτει και την ε, ευαισθησία του δέρματος, όπως επίσης και την πρόκληση καρκίνου. Αυτά για την απαγόρευση του 2013. Και απορρέουν όλα αυτά από τα συμπεράσματα της ομάδας. Δεν υπήρξε αντίρρηση, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και επιβεβαιώθηκε η κατάσταση αυτή πολλές φορές μάλιστα από την Επιστημονική Επιτροπή για καταναλωτικά προϊόντα και πιο πρόσφατα από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια Καταναλωτών. Όλα αυτά για την τοξικότητα σε επανελειμμένη δόση. Ενημερώθηκε σχετικά και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την έκθεση του 2005 και του 2006, αλλά και με απαντήσεις που στείλαμε σε γραπτές σας ερωτήσεις. Η επανελειμμένη αυτή δόση αναφέρεται πολλές φορές και στην οδηγία για τα καλλιτικά και χρησιμοποιείται για να καλύψει διάφορες κατηγορίες τοξικότητας που εμφανίζονται μετά από επανειλημμένη έκθεση στα προϊόντα. Σήμερα λοιπόν βάσει τις οδηγίες καλλιτικών η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2011 για τις εξελίξεις και για την έγκριση εναλλακτικών μεθόδων, ιδιαίτερα για τα σημεία που έχουν να κάνουν με την απαγόρευση του 2013. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν την κατάσταση, φτιάξαμε ομάδες εμπειρογνωμόνων, όπου συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Ορίστηκαν όχι ως εκπρόσωποι κάποιας ε, πλευράς, αλλά ως άτομα ο κ. Μπεζέ προεδρεύει και ετοιμάζουν ένα σχέδιο τεχνικής έκθεσης. Αυτή η τεχνική έκθεση έχει ως στόχο να απεικονίσει όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και πλήρως τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που διαθέτουμε για την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων όσον αφορά τα, τις απαγορεύσεις που προβλέπονται για το 2013. Προβλέπει έκθεση επίσης και αξιολόγηση βάσει επιστημονικών δεδομένων για το χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση των ε, πειραμάτων με ζώα. Τώρα γίνεται διαβούλευση, μάλλον ολοκληρώθηκε μόλις και η τεχνική αυτή έκθεση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Βάσει αυτής της τεχνικής έκθεση, λοιπόν η Επιτροπή θα ετοιμάσει και την επόμενη έκθεσή τη που θα στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Συγχρόνως θα κάνουμε μια ανάλυση αντικτύπου για να ετοιμάσουμε την ε, απόφαση που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την προθεσμία του 2013. Για τα σημεία που καλύπτονται από την ημερομηνία αυτή, η οδηγία καλλιντικά προβλέπει την δυνατότητα να κάνει νομοθετική πρόταση η Επιτροπή στην περίπτωση που εναλλακτικέ μέθοδοι δεν έχουν αναπτυχθεί ή δεν έχουν εγκριθεί μέχρι το 2013. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα υπάρξει πρόταση και αν ναι, τι θα περιλαμβάνει. Η ανάλυση αντικτύπου λοιπόν θα μας επιτρέψει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες των διάφορων αναλλακτικών λύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κατριν Σουλία τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η τεχνική έκθεση περίφημη που μόλις ακούσαμε, θέλω να ξέρω η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας, Επιτροπή Περιβάλλοντος και πότε, εάν η απάντηση είναι καταφατική. Ο Κρις Ντέβης. Ομολογώ ότι εκπλήσαμε που μου δώσετε λόγο πριν από την κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ε, γιατί η Ντάκμαρ ήταν η συγγήτρια όταν ε, ετέθη το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να κάνω απλά κάποιες ερωτήσεις. Φτάσαμε λοιπόν ε, στην καταληκτική ημερομηνία και ποια είναι η εναλλακτική λύση. Ποια είναι η αξιολόγηση του πότε θα καταστεί δυνατόν να αντικαταστήσουμε ε, τις, ε, ε, τα πειράματα στα ζώα με πειράματα που δεν θα περιλαμβάνουν ζώα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το ότι προκαλούμε πόνο στα ζώα για να παραχθούν νέα προϊόντα. Ενώ κατ' ουσίαν ε, αυτό που θέλουμε είναι να ε, βελτιώσουμε την ανθρώπινη εμφάνιση. Δεν μιλάμε μόνο για το make-up ε, και τα καλλιτικά, μιλάμε και για προϊόντα ατελείωτα προϊόντα μπάνιου. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδων make-up και πολλά πολλά άλλα καλλιτικά. Το θέμα είναι, μα επιτέλους δεν μπορεί ο ανθρώπινος πολιτισμός να ε, προχωρήσει για την επόμενη δεκαετία χωρίς να γίνουν άλλα πειράματα για τέτοιου είδους προϊόντα. Όλη αυτή η στρατηγική βασίζεται στην ιδέα του να υπάρχουν νέα προϊόντα ε, τα οποία θα ε, προσφέρονται τα Χριστούγεννα στα γενέθλια και ότι αν δεν συνεχιστεί αυτό υποτίθεται θα καταρρεύσει ο κλάδος. Όμως ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς έχει αξιολογήσει τις ε, επιπτώσεις στην απασχόληση. Θα πούμε ή δεχόμαστε απλά ότι ο νόμος είναι αυτός που είναι και η τελικά η θα τεθεί σε ισχύ όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. Ευχαριστώ, Κρυ. Η ε, Ντάκμαρ τώρα. Ζητώ συγγνώμη κιόλα. Δεν χρειάζεται να ε, ζητάτε συγγνώμη. Ε, δεν χρειάζεται να τα υποθέτετε αυτά αυτομάτως επειδή μιλάμε για καλλιντικά. Ε, κάπου στη δεκαετία του 90 έγινε η έκτη αναθεώρηση, τώρα γίνεται η έβδομη αναθεώρηση του ίδιου νομοθετήματος. Ε, πολλοί συνάδελφοι ήταν μέχρι τις 3.30 το πρωί στη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν ότι η αναχείρας νομοθεσία ήταν ε, ε, καλή αλλά και δύσκολη. Και η τελευταία το ίδιο. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια προς τη Δεπιαν Λεγκρενιέ και προς τη Γάμα Δέλτα Σάνκο, έτσι, που, την οποία εκπροσωπεί. ό,τι και να γράφετε στις εκθέσεις σας, ό,τι και αν διαφύγει της προσοχής μας την επιστολή, κοιτάξτε, είμαστε αντιμέτωποι με την νομοθεσία. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Τι λέει λοιπόν η νομοθεσία. Στο άρθρο 4, α 2.1 μάλλον, για τις ε, δοκιμές ε, τοξικότητας, ε, τοξικότητας για την αναπαραγωγή ε, δεν λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή της παραγράφου 1 και περιοριζόμαστε κατά το όριο στα 10 χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας. Ε, το 2013 όμως συζητάμε τώρα, ε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, μιλάμε για τρεις διαφορετικές δοκιμές και δεν μιλάμε για καρκινογόνες ουσίες και δεν μιλάμε για ευαισθητοποίηση του δέρματος. Το τελευταίο θέμα με ενοχλεί ακόμη περισσότερο. Για ε, τα τεστ στο δέρμα δεν μπορώ καν να το προφέρω. Ε, θα πρέπει να ε, κάνω πρόβες. Τα ίδια είχα πάθει και με τις εγκεφαλοπάθειες. Πριν από 15 χρόνια λοιπόν ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα χρειαζόμασταν πλέον δοκιμές σε ζώα. Είπε ναι και η βιομηχανία και όσοι δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με το θέμα Καμία δοκιμή για τα καλλιντικά ποτέ δεν εγκρίθηκε. Δεν μπορεί η δοκιμή με τα ζώα να είναι συγκρίσιμη με τη δοκιμή σε ανθρώπους. Άλλο όταν μιλάμε για λαγούς, για ε, κουνέλια, για ποντίκια, ε, για ρουρέους. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν κάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, για τις ε, ε, καρκινογόνες ουσίες και ε, για την ευαισθητοποίηση του δέρματος, συμφωνούμε ότι δεν θα ισχύσει η ημερομηνία το 2009 και θα συνεχιστούν μέχρι το 2013 οι δοκιμέ. Αυτό είναι το πρώτο. Ε, εκνευρίστηκα λίγο, ή μάλλον να το πω καλύτερα, εξεπλάγιν, από την ειλικρίνειά σας. Ήρθατε και μας είπατε και αναρωτηθήκατε τι θα γίνει αν δεν έχουμε εναλλακτικέ ε, λύσεις για τις καρκινογόνε ε, ουσίες, ε, για την αναπαραγωγική τοξικότητα επίσης η Φρανσουάζο, ο Κρίς, οι συνάδελφοι που ήταν τότε σε αυτή τη συνδιαλλαγή που σας έλεγα προηγουμένως, το ξέρουν. Η βιομηχανία μας είπε τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα έχουμε συγκεκριμένα αποτέλεσμα. Και είπαμε εμείς εντάξει θα χορηγήσουμε εξαίρεση. Δεν ε, το καταλογίζω στη βιομηχανία. Υπήρχε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τη Βιομηχανία. Ε, ό,τι και να έγινε πάντως δεν επαρκεί. Σαμπίν δεν συμφωνώ όμως να εξετάζουμε τώρα μέτρα για να επιμηκύνουμε την ε, προθεσμία. Αν αρχίσουμε τώρα το 2013, όπου θα υποβάλλεται πρόταση νομοθετήματος που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για συναπόφαση, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει, θα σας πω ότι εγώ σίγουρα δεν θα είμαι συγγήτρια τότε. Αλλά το 2014 πριν τι εκλογέ, θα φέρετε κάτι τέτοιο εδώ στο Κοινοβούλιο. 20 χρόνια και δηλαδή θα το συζητάμε τότε. Και θα έχουμε τα ίδια επιχειρήματα που μόλις ακούσαμε από τον Κρίς. Ε, δεν σε κατακρίνω τώρα. 15 χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια τα ίδια λέγαμε. Δίκιο έχετε, αλλά ε, λίγους μήνες πριν τις εκλογές θα αρχίσουμε να τα ζητάμε αυτά στο Κοινοβούλιο για την ευημερία των ζωών. Ξέρετε τι, θα ασφαχτούμε και θα έχουμε πολλά μικρά κομματάκια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Διάβασα με προσοχή την εκθεσή σας. Διάβασα αυτά που είπατε, σελίδα 4, όχι 4, 8, τις πληροφορίες προς τα κράτη-μέλη, πολύ ωραία αυτά. Όλα τα διάβασα. σαφέστατα όμως για τις ε, δοκιμές, ούτε καν να το σκεφτείτε. Πρέπει, ε, κανονικά έπρεπε σταδιακά να έχουν ήδη καταργηθεί, ήδη από πέρσι. Πω, δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε αλλιώς την νομοθεσία προσέξτε αν αλλάξετε ε, την 7η αναθεώρηση με την προθεσμία του 2013. Ξέρετε τι θα γίνει, όλοι το γνωρίζουν τι θα γίνει. Ένα πράγμα, για κάθε νέα ενεργό, ε, ενεργή ουσία δεν είναι και τόσες πολλές. Ε, γιατί μία δοντόκρυμα που ασπρίζει τα δόντια, λευκένει τα δόντια. Για ένα νέο αποσμητικό που χάρη στο οποίο δεν θα υδρώνουμε όχι για 24 ώρες, για ολόκληρη τη βδομάδα. Δεν γίνεται με, τα νέα προϊόντα. Δεν γίνεται να αδειοδοτηθεί αυτό το προϊόν άμα έχουν γίνει δοκιμές με ζώα. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης στην αγορά. Και πολύ αμφιβάλλω αν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις μια νέα αναθεώρηση. Τα έχουμε δοκιμάσει ήδη. Ε, στο παρελθόν όλα, όλες τις ουσίες ε, ε, ε που χρησιμοποιούνται για τα καλλιντικά. θα πρέπει να, να το πούμε ομά. Δεν ενδιαφέρεται κανεί αν θα ειναι Απρίλιος, Μάιος. Πάντως, 2013 θα είναι. Και μην ξεχνάτε τις πολιτικές επιπτώσεις. Εγώ ήδη παίρνω επιστολές. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι, αλλά Όσοι δεν είναι εδώ και τόσα χρόνια όπως εγώ στο Κοινοβούλιο, να σας πω ότι πραγματικά ε, με την πρώτη πρόταση και τη δεύτερη ε, πήρα πάνω από 24.000 πάνω από 24.000 επιστολές στο σπίτι μου σε ένα τόσο δα γραμματοκιβώτιο. Ε, τέσσερις με έξι μήνες πριν εγκριθεί η νομοθεσία. Με μίσησε ο ταχυδρόμος. Η βιομηχανία είχε δεχτεί την προθεσμία, είπανε ωραία πολύ γενναιόδοροι είσαστε που μας δίνετε ε, και άλλα χρόνια για, για, την, καρ... για τις καρκινογόνες ουσίες ε, και για την τοξικότητα. Αυτά. Merci beaucoup. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ εκ μέρους της ομάδας μου για τις παρατηρήσεις ε, της εισηγήτριας. Μην παρετηθούμε, μην κάνουμε πίσω. Σίγουρα θα πετύχουμε ειδική πλειοψηφία. Και θα τηρηθούν οι προθεσμίες. Όσον αφορά τώρα τα επιστημονικά πειράματα στα ζώα, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη υγεία, τότε αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν όμως πράγματα, όπως είναι τα καλλιντικά, που δεν χρειάζονται πειράματα σε ζώα. Συμφωνώ λοιπόν και να τηρηθούν οι ημερομηνίε και όλα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα που είναι ανθρώπινη υγεία και αυτό επιμένω είναι διαφορετικό. Για μας είναι αναγκαίο να γίνονται αυτά που γίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον. Συμφωνώ με την εισηγήτρια για το ότι πρέπει να υιοθετήσουμε στάση που αν τροποποιεί την ήδη υπάρχουσα θέση θα γεμίσουμε από καινούρια γράμματα. Να ξέρετε ότι όλοι μας έχουμε πάρει ακόμα και υβριστικά μηνύματα όταν αλλάξαμε τις θέσεις μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για καλλιτικά και για προϊόντα που δεν σώζουν ανθρώπινες ζωές, τα πράγματα είναι αλλιώς. Οι προθεσμίες δεν πρέπει να τροποποιηθούν, όπως λέει και η συγγήτρια. Συμφωνώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Φιλίπ Πρόεδρε, υπάρχουν δύο προτεραιότητες ε, που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Η πρώτη για όλου, προτεραιότητα για όλους, είναι ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια για του καταναλωτέ. Αυτό είναι η ψηστή προτεραιότητα. Ε, δεν μπορούμε να περιέχουμε στην εξή κατάσταση ότι επειδή επιβλήθηκε εναλλακτική μέθοδος παρότι δεν την ελέγχαμε πλήρως τελικά διατέθη στην αγορά ένα προϊόν που ε, απεδείχθη επικίνδυνο. Οι εναλλακτικέ ε, μέθοδοι τώρα εκπονούνται. Γνωρίζουμε όμως σήμερα ότι δεν είναι τελειοποιημένες είναι δύσκολο κατά τη γνώμη μου να πούμε ότι θα τηρήσουμε την προθεσμία γιατί έτσι το υποσχεθήκαμε ενώ ε, στην ε, πράξη δεν είναι έτοιμες οι μεθοδολογίες. Ποιο θα πάει ενώπιον των καταναλωτών δηλαδή και θα του πει ότι ε, έχουμε μία λίγο χειρότερη μέθοδο αξιολόγηση, αλλά αποφασίζουμε να την εφαρμόσουμε γι' αυτό γι' αυτό τον λόγο. Λοιπόν, ε, ύψιστη προτεραιότητα η υγεία του καταναλωτή. Έχει θεμελιώδη σημασία. Κατόπιν. οι δοκιμές in vivo και in vitro με τα ζώα δεν μας δίνουν τα σωστά στοιχεία μας λέτε σε σχέση με αυτά που γίνονται με τις δοκιμές σε ανθρώπους. Εξαρτάται, εξαρτάται. Αν μιλάμε για καλλιτικά, αν μιλάμε για φάρμακα, οι δοκιμές, οι εργαστηριακές δοκιμές μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε τα όσα ισχύουν για τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν έχουμε ανασυνθέσει ανθρώπινο δέρμα σε εργαστήριο, αυτό είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον. Δηλαδή, μπορούμε κάποια στιγμή να αφήσουμε τις παλιέ ε, μεθόδους δοκιμής. Αλλά ε, οι σημερινέ μέθοδοι ανασύνθεσης ε, ε, του ανθρωπίνου δέρματος δεν είναι τελειοποιημένε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή υποσχεθήκαμε μία προθεσμία, αντί και καλά πρέπει να την εφαρμόζουμε, προσβάλλοντας την υγεία του καταναλωτή. Δεύτερον, πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι. Η βιομηχανία των νοκαλυτικών είναι μια ανθυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και άρα είναι πηγή πλούτου ε, για την Ένωση με τέτοιους, λοιπόν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυστηρούς κανόνες και να αποθέσουμε ένα μεγάλο άχθος σε αυτή τη βιομηχανία, ε, να βαρύνουμε αυτή την βιομηχανία, ε, ενώ σήμερα ε, στα ε, καλλιντικά ανθίζει αυτή η βιομηχανία, έτσι θα εκτοπιστούν οι βιομηχανίες από την Ευρώπη. αντί να χοροπηδάμε και να λέμε όχι, όχι, εγώ θέλω το 2013, το 2013, το 2013, ε, όχι, πρέπει να συνυπολογίσουμε αυτά τα στοιχεία. Προστασία του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, προστασία της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, που δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με όλες αυτές τις ε, δυσκολίες και ε, προ όφελο άλλων βιομηχάνων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα χρειαστεί να συμμορφωθούμε του ίδιου κανόνε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ε, μου ξαναδώσατε το λόγο ε, και ζητώ συγγνώμη που ξαναπήρα το λόγο πριν από τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους. Εδώ πραγματευόμαστε μία νομοθεσία που είναι υποχρεωτική. Στην Γαλλία, αν είσαι αυτή η νομοθεσία, μπορείτε να προσπαθήσετε ε, όλοι να την τροποποιήσετε, αλλά ε, τον των, κανόνων που ισχύουν στη Γαλλία. Τώρα όμως εδώ στο Κοινοβούλιο, για να υπάρξει τροποποίηση, χρειάζεται πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω πώς θα ήταν αυτό εφικτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ καν πόσες συνεδριάσει, συναντησει συγγνώμη, είχαμε εκπροσώπους της ΛΟΡΕΑΛ. Πάρα πολλε Η ΛΟΡΕΑΛ είχε πολύ ε, ισορροπημένη ε, στάση και το ίδιο και ο Ευρωπαϊκός ε, Αρμόδιος Οργανισμός. Ε, για τις ε, λοιπές εναλλακτικέ μεθόδους, ε, για τις δοκιμές in vitro, τα θέματα της σήμανσης, Το θέμα είναι περίπλοκο. Εξαρτάται ο καθένας από ποιους εκλέγεται, από ποια χώρα εκλέγεται και σε ποιους, και ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται προς όφελος των καταναλωτών. Εδώ και 21 χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και μάχομαι για την προστασία των καταναλωτών. Ποιος θα έρθει εμένα να μου ε, δώσει να μου, ε, μαθήματα σχετικά με το πώς θα προστατεύω τους καταναλωτές. Όπως και για τα τσιγάρα, έτσι και στα καλλιτικά μπορούμε να πούμε έγινε ε, δοκιμή σε ζώα και ας αποφασίσει ο καταναλωτής αν θέλει να ε, χρησιμοποιήσει αυτά τα καλλιτικά. Στα τρία τέταρτα των χωρών, ξέρετε ποια θα είναι η αντίδραση, δεν θα αγοράσει κανεί αυτό το προϊόν. Ε, έχετε εκατοντάδες ήδη οδοντόκρεμας στα καταστήματα. Και αν 10 έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, ε, λοιπόν θα πάει, ε, θα πάει ο καταναλωτή και θα αγοράσει κάτι άλλο. Η, η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών δεν θα αγοράσει μια οδοντόκρεμα που έχει δοκιμαστεί σε ε, ζώα. Τώρα, η ευρωπαϊκή και η διεθνή ε, βιομηχανία. Εγώ εδώ και 20 χρόνια ε, συνομιλώ με την CTFA που είναι η ε, συνομοσπονδία των Αμερικανικών βιομηχανιών. Η νομοθεσία που ψηφίζουμε εδώ επηρεάζει ε, και την Κλινή και την Εστελόντερ και τη Λορεάλ ανά τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια περίοδο ανώ των 18 μηνών, πρέπει να φέρει σήμαση ημερομηνία λήξης. Εάν έχει μακρύ ε, κύκλο ζωής ε, το προϊόν, ε, θα πρέπει να φέρει αυτό το εικονίδιο, ε, μία κρέμα με ανοιχτή, με ένα δάχτυλο μέσα που θα γράφει 6, 9, 12 μήνες. Για πόσους μήνες δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν από τη στιγμή που θα ανοιχθεί. Οι Αμερικανοί ε, διαφώνησαν μαζί μου για πάνω από ένα χρόνο, γιατί γνωρίζουν πως η νομοθεσία που εγκρίνουμε εδώ θα εφαρμοστεί λιγάκι σε αυτούς. Άρα τα όσα αποφασίζουμε εδώ δεν επηρεάζουν μόνο την Ευρώπη, είτε μιλάμε για το περιβάλλον, για τα τρόφιμα, οτιδήποτε. Δεν επηρεάζει μόνο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αλλιώς, ας κάτσω εγώ στο Βερολίνο, καθίστε εσείς στη Γαλλία λοιπά. Δεν μπορούμε να έχουμε εναλλακτικέ προαιρετικέ νομοθεσίες. Όταν έχετε την 7η αναθεώρηση της οδηγίας για τα καλλιτικά, ε, συγγνώμη, έχει εγκριθεί, ισχύει και δεν μιλώ ως δικηγόρος αλλά ως νομοθέτης. Είναι δεσμευτική, δεσμευτικό το νομοθέτημα αυτό. Πρέπει να το τηρήσουμε και προβλέπεται προθεσμία και πρέπει να τηρηθεί γιατί είναι νόμος. Αν θέλετε να αλλάξουμε την νομοθεσία, όπω είπε η κυρία Λεγκρινιέ, πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία. Άρα χρειαζόμαστε νέα πρόταση. Ε, πρέπει να περάσει από δύο αναγνώσει, είναι διαδικασία συναπόφαση Ε, πρέπει να περάσουμε από τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία όπω λέγεται τώρα αλλά πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, θα κάνω να το σκέφτεστε. Ε, Α σκεφτούμε μια άλλη λύση που να μην συνεπάγεται ε, τροποποίηση τη νομοθεσία. Η κυρία yeah. Πολύ σύντομα και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση δείχνει ότι εδώ είμαστε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Η προστασία του καταναλωτή, όπως λέει και ο κύριος Ζωβάν, αλλά και η προστασία των ζώων. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Μην μεταφέρουμε τα πειράματα στα ζώα σε άλλες χώρες, όπου εκεί σέβονται πολύ λιγότερο τα ζώα από ότι εμείς. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία, πράγμα το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές. Κύριε Ζουβά, μακριβώς θέλω να απαντήσω στη συνάδελφο. Είναι ένα περίπλοκο θέμα και εγώ θέλω να το δω με ρεαλισμό και όχι ιδεολογικά. Υπενθυμίσατε ότι είστε νομικός και ευρωβουλευτής. Εγώ είμαι γιατρός και ευρωβουλευτής. Εντάξει, μπορεί να βλέπω τα πράγματα λιγότερο από την νομική άποψη, αλλά ανησυχώ, δεν λέω ότι πρέπει να ανησυχούμε, αλλά τόσο πάντων με απασχολεί περισσότερο η ιατρική, επιστημονική πλευρά εφαρμογή των πειραμάτων στα ζώα. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι θέλουμε, αν όταν το αποφασίσουμε το 2013, αν είναι το 2013, δεν έχουμε εναλλακτικέ δοκιμές, ε, δεν θα έχουμε. Μπορεί να φωνάζουμε και να λέμε να έχουμε, να έχουμε, να έχουμε, αλλά τότε τι θα γίνει, εφόσον υπάρχει απαγόρευση, θα γίνονται αλλού τα πειράματα. Και θα είναι σε βάρο τη δικιά μα ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν ζούμε σε ένα κόσμο ιδανικά πλασμένο. Όχι, φυσικά, μακάρι να αντικατασταθούν όλα τα πειράματα. Αλλά αν δεν έχουμε εναλλακτικέ μεθόδους, ξέρουμε τι μας περιμένει. Ο κύριος Περλάτο. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να καλέσω τους συναντέλφου ε, να ε, είναι συνεπείς σε αυτό που θα μπορούν να αποβούν συνέπειες ε, των επιπτώσεων και να δείξουν ότι γνωρίζουν τις συνέπειες αυτές η εφαρμογή της απαγόρευσης ε, προφανώς ε, θα ε, συνεπάγεται την μετεγκατάσταση, τη μεταφορά των πειραμάτων σε άλλες χώρες. Κατόπιν τούτου είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε πρώτα απ' όλα την υγεία των πολιτών, των ανθρώπινων όντων. Βέβαια <clears throat> πρέπει να δώσουμε και μία απάντηση σε αυτή την αυξανόμενη ευαισθησία όσον αφορά ε, το σεβασμό των ζώων. <clears throat> Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τους ισχυρισμούς μας, το να διατηρηθεί η απαγόρευση των πειραμάτων όσον αφορά τα καλλιντικά, γιατί πρέπει να προσέξουμε ακόμα και τα καλλιντικά ε, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην ανθρώπινη υγεία. Μπορούν να είναι και καρκινογενή. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν να πούμε εντάξει απαγορεύονται καλλιντικά και για να δώσουμε μία απάντηση στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση δεν πρέπει να απαγορεύσουμε μόνο τις, τα πειράματα σε ζώα αλλά και το, τη χρήση την εμπορευματοποίηση, την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ε, πειράματα σε ζώα σε άλλες ε, περιοχές και βιομηχανίε εκτός Ευρώπης. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει να απαγορεύσουμε τα πειράματα στην Ευρώπη και όπως συμβαίνει και με άλλες, ε, άλλα προϊόντα να επιτρέψουμε την εισαγωγή προϊόντων που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου, από χώρες όπου γίνονται αυτά τα πειράματα. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Το δεύτερο, κοιτάξτε, ε, επειδή αυτά συμβαίνουν, είμαστε αναγκασμένοι, οι βιομηχανίες μας είναι αναγκασμένες να ανταγωνίζονται και εδώ πάω πιο πέρα από τα καλλιτικά. Είναι λοιπόν αναγκασμένες οι βιομηχανίες μας να ανταγωνίζονται στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Είναι αναγκασμένες λοιπόν οι βιομηχανίες μας να ανταγωνίζονται με χώρες που δεν εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει η Ευρώπη. Ούτε έχουν και τον ίδιο σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ούτε και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον. Και μάλιστα τα προϊόντα τους ε, τα φέρνουν εδώ και κάνουν ε, παράνομο, αθέμητο ανταγωνισμό και με τον τρόπο αυτό οδηγούν ε, στην εξαφάνιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αν λοιπόν θέλουμε να ενστερνιστούμε αυτή την υπόθεση, δηλαδή της ε, προστασίας των ζώων, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να πάμε πιο πέρα, όχι απλά να απαγορεύσουμε τα πειράματα στην Ευρώπη, αλλά να απαγορεύσουμε να ε, ε, εισάγουν στην Ευρώπη προϊόντα από άλλα μέρη του κόσμου και μάλιστα με πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Αξίζει την προσοχή μας. Και ανησυχώ όχι μόνο για τα μήλα, γιατί ε, είχαμε κάποια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, κάποια αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τα ζώα που ε, χρησιμοποιούνται για πειράματα. Και απ' την άλλη κάποιοι ζήτησαν την ε, απελευθέρωση των πειραμάτων σε ζώα. Κάτι που είναι τελείως λάθος. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από λίγους που είναι όμως οργανωμένοι και θέλουν να δείξουν ότι είναι εκατομμύρια απειλώντας μας ε, να μας δολοφονήσουν εμάς και τους συγγενείς μας, κάτι το οποίο θεωρώ παντελώς απαράδεκτο. Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα αντικειμενικά, θα πρέπει να αποφασίσουμε αγνώντας τους συναισθηματισμούς. Νομίζω και ελπίζω ότι το θέμα αυτό θα το εξτάσουμε με απόλυτη νυφαλιότητα. Βεβαίως και να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, ανθρώπινη ζωή, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση όσον αφορά αυτή την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση που αφορά στην προστασία των ζώων. Κριστέβης και μετά θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να παρεύω και πάλι. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι υπάρχει πλήρης απαγόρευση καλλιντικών μετά από... Ε, για πειράματα στα καλλιντικά. Μα εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο για αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, μας ενδιαφέρει και το ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλουμε τέτοια καλλιντικά. Θυμάμαι το 97 και 98 που είχαμε τη νέα εργατική κυβέρνηση στο Ενωμένο Βασίλειο τότε και ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε ήταν να απαγορεύσουν στο Ενωμένο Βασίλειο τα πειράματα σε ζώα καλλιτικά. Ε, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνα στη Γαλλία και κάνα τα πειράματα. Εντάξει, δεν το λέω τώρα αντίον των Γάλλων. Θέλω να πω. Αν λοιπόν θέλεις σοβαρά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σιγά σιγά και πιο πέρα. Με προθεσμίες να φροντίσεις να έχεις μια πλήρη απαγόρευση στην αγορά των καλλιντικών. Πλήρη. Τώρα, όσοι από εσά είστε πιο πρόσφατοι, δεν θα ξέρετε ότι υπάρχουν ε, κάποιε εταιρείε καλλιντικών που δεν έχουν ιδέα για το τι σκέφτεται ο κόσμος για αυτά. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ την τελευταία δεκαετία, η αντιμετώπιση του δηλαδή. Η βιομηχανία έχει συνεργαστεί με τις κυβερνητικές οργανώσεις, με επιστήμονες κτλ. Υπάρχει μια αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν προχωρήσει με την παραγωγή καλλιτικών που δεν χρειάζονται πειράματα στα ζώα. Βέβαια, πάντα ξέραμε ότι κάποια πειράματα θα ήταν δύσκολο να αντικατασταθούν. Να βρεθούν άλλες λύσεις, να μην είναι πειράματα σε ζώα. Τώρα, μας θυμίζει η Επιτροπή, πλησιάζει η προθεσμία. Τώρα εγώ εδώ θα συμφωνήσω με την Τάκμα Μπένετ. Μερικοί θα πούν, ναι, το ξέραμε. Αλλά επιμένουμε ότι μετά το 2013 δεν θα επιτρέπουμε νέα καλλιντικά εφόσον έχουν γίνει πειράματα για αυτά σε ζώα. Η εναλλακτική λύση ποια θα είναι. Ίσως να πούμε θα επιτρέψουμε νέα προϊόντα, αλλά να λένε απάνω τα προϊόντα σας αυτά, εφόσον έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, ότι για να φτιαχτούν αυτά τα καλλιντικά έχουν γίνει πειράματα σε ζώα, με μεγάλα γράμματα. Και τότε να δούμε τι θα πούνε. Γιατί τότε οι καταναλωτές θα το βλέπουν πάνω στο προϊόν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματόζωα για αυτά και θα είναι δικιά τους επιλογή τι θα κάνουν, θα τα αγοράσουν ή όχι. Έχουμε καλή νομοθεσία προς το παρόν, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικέ λύσεις αντί για πειράματα στα ζώα. Γι' αυτό θέλω να μου πει η Επιτροπή. Στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, εγκεκριμένες. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απαγόρευση. Πρόεδρος, ήρθε και η κυρία Όγκο, οπότε θα μπορέσουμε να δούμε και το προηγούμενο σημείο. Κύριε Γνενιέ, για να προχωράμε λίγο-λίγο. Για απαντήστε παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την τεχνική έκθεση, που πρέπει να δείχνει ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά εναλλακτικέ μεθόδους, αντί για πειράματα. Η τεχνική αυτή έκθεση έγινε για να παρουσιάσει μια πιο πλήρη και ουδέτερη εικόνα της κατάστασης γίνεται. Και γι' αυτό και την αναθέσαμε σε πυρογνώμονε από τι κυβερνήσει, από τη βιομηχανία, από την ΕΚΒΑΜΑ, από την Επιστημονική Επιτροπή και από ομάδε προστασία των ζώων, ώστε όλοι μαζί να εκπονήσουν το σχέδιο έκθεσης. Αυτό το σχέδιο ε, περνάει από διαβούλευση. Θα δούμε τι σχόλια θα έχουν γίνει και θα ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, στα τέλη της χρονιάς. Ποια είναι τα προσωρινά αποτελέσματα από την έκθεση αυτή. Αν δούμε ένα χρονοδιάγραμμα για να δούμε πόσο γρήγορα προχωράμε σε εναλλακτικέ μεθόδους αντί για πειράματα σε ζώα. Για την ε, ευαισθησία του δέρματος για το 2007-2019 μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές μεθόδους. Για την τοξικό κινητικότητα, 5 με 7 χρόνια για να έχουμε εναλλακτικέ μεθόδους. Για την αναπαραγωγική τοξικότητα, 10 χρόνια περίπου. Και για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις τοξικότητα, και δημιουργία καρκίνου, οι εμπειρογνώμονε δεν μπόρεσαν να πούνε σε πόσο χρόνο θα έχουμε εναλλακτικέ μεθόδου. Αυτά είναι τα τεχνικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα και που απορρέουν από όλου αυτού του εμπειρογνώμονε. Σα είπα, θα χτενιστεί ακόμα η έκθεση, θα ληφθούν υπόψη και τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση. Και εννοείται μπορούμε να έρθουμε και να σα παρουσιάσουμε εδώ την έκθεση αυτή όταν θα έχει ολοκληρωθεί. Ποια είναι τώρα η νομική κατάσταση. Όπως είπαμε, δεν συζητάμε τώρα τη δυνατότητα να κάνουμε πειράματα μέσα στην Ευρώπη με ζώα για τα καλλιντικά. Από το 2009 το έχουμε πει αυτό, οπότε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται πια τέτοια πειράματα για καλλιντικά. Αυτό που συζητιέται τώρα είναι θα επιτρέπεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορία προϊόντων τα οποία έχουν δοκιμαστεί πάνω σε ζώα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το μεγαλύτερο μέρος των πειραμάτων η απάντηση είναι αρνητική. Όχι. Αλλά υπάρχουν ακόμη τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση από το 2013 και μετά. Όσον αφορά λοιπόν την εμπορία και μόνο για αυτές τις κατηγορίες η οδηγία αφήνει μια πόρτα ανοιχτή λέγοντας ότι εάν διαπιστώσουμε το 2011 ότι δεν έχουμε εναλλακτικέ μεθόδους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τότε να κάνει πρόταση. Πρόταση η οποία εφόσον γίνει θα πρέπει να εγκριθεί με συναπόφαση. Αν λοιπόν πρέπει να κάνουμε πρόταση θα την κάνουμε το 2011 ώστε να εγκριθεί με συναπόφαση το 2013. Ακόμα δεν έχουμε πάρει καμιά απόφαση Ετοιμάζουμε μια ανάλυση αντικτύπου όμως που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πλευρές του ζητήματος. Την προστασία των ζώων, πόσα ζώα χρησιμοποιούνται ή επίσης πόσο έχουμε προχωρήσει στις ερευνητικές προσπάθειες για εναλλακτικέ λύσεις. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη μας την ασφάλεια του καταναλωτή και την, όταν μιλάμε για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, γιατί για ορισμένε ουσίε που κυκλοφορούν σήμερα ω καλλιντικά, επειδή η επιστήμη εξελίσσεται, πρέπει να γίνουν ξανά πειράματα, να δοκιμαστούν αυτέ οι ουσίε. Και τι βαφέ για τα μαλλιά, για παράδειγμα, έχουν γίνει δοκιμέ στα ζώα. Ξανά. Πρέπει να δούμε επίσης και τις συνέπειες που απορρέουν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Να δούμε τις συνέπειες στην απασχόληση, στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και στο εμπόριο, γιατί όπως είπαμε είναι μια κατάσταση που επηρεάζει πολύ και την θέση μας στην διεθνή εμπορική σκηνή. Αξιολογώντας λοιπόν τον αντίκτυπο όλων αυτών, έχουμε μια συγκεκριμένη γνώση των συνεπειών των αποφάσεων που θα πάρουμε. Όποιες και αν είναι αυτές. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά όποια και αν είναι η απόφαση που θα πάρουμε, θα ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες, οπότε θα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και τις ευθύνε μας για αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα έτσι κι αλλιώς, του χρόνου δίχως άλλο. Προτείνω τώρα να περάσουμε στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που ήταν το σημείο 8 έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων την αντινήσπραξη τελών. Το λόγο έχει πρώτο ο κύριο Μπερνάρ ο οποίος είναι ε, στην ΣΑΝΚΟ, γενικός στη ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω την έκθεση που ενέκρινε τον προηγούμενο μήνα η Κομισιόν και έχει σχέση με, τις, ε, με την ίσπραξη τελών στην Ευρωπαϊκή Αρχή ασφάλεια Τροφίμων. Αυτή η αρχή είναι πολύ σημαντική για όλους μας, ε, κυρίως για σας. Γι' αυτό λοιπόν και η έκθεση αυτή ε, είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να ομολογήσω ότι την έκθεση αυτή πρέπει να την έχουμε καταθέσει πριν από πέντε χρόνια, αλλά τότε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Χρειαζόμασταν χρόνο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή να ε, λειτουργήσει εύρυθμα και να γίνουν κατανοητές οι δραστηριότητες της. Από τότε που συστήθηκε η αρχή αυτή ε, προσθέθηκαν πόροι γιατί η χρηματοδότησή της ανέλαβε περισσότερες ευθύνες. Έτσι λοιπόν χρειαζόμασταν και περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουμε ακριβώς ε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το θέμα των τελών προς την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας ε, Τροφίμων. Έπρεπε να ληφθεί υπόψη ο νέος κανονισμός που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Αυτή Αρχή, την ΕΦΣΑ και η εμπειρία μας έδειξε ότι οι φάκελοι που κατατίθενται από τους ετούντες δεν είναι πάντα ικανοποιητικοί. Η ΕΦΣΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή ε, ασφάλεια τροφίμων, τώρα πλέον βρίσκεται σε μια φάση σταθεροποίησης. Για να έχετε έτσι μια εικόνα, η επεξεργασία ε, θεμάτων από την ΕΦΣΑ αποτελεί τώρα το 31% του προπολογισμού, ενώ πριν από τρία χρόνια το ποσοστό αυτό ανήρχεται σε 15%. Είναι λοιπόν σκόπιμο και φυκτό να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα ε, τελών υπέρ της ΕΦΣΑ. Και εδώ ε, συμβουλευτήκαμε όχι μόνο την ΕΦΣΑ αλλά και τα κρατημέλη και τους άμεσα ενδιαφερόμενους για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το θέμα. Και το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο από αυτού γιατί νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να το συζητήσουμε το θέμα. Το βασικό λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι είναι πολύ περίπλοκο το να υπάρχει ένα ε, σύστημα εισπραξής τελών στον τομέα της ε, νομοθεσία τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο ε, και να καταλήξουμε τελικά σε μελέτη επιπτώσεων. Στη δική μας την έκθεση εντοπίζουμε τέσσερις εναλλακτικέ λύσεις που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Η πρώτη αφορά σε ένα εφάπαξ ποσό για όλες τις αδειοδοτήσεις. Η δεύτερη εναλλακτική αφορά τέλη για όλες τις αδειοδοτήσεις. Τρίτη εναλλακτική τέλος, όπου το τέλος αυτό ποικίλει ανάλογα με τον ε, τούντα, με την ουσία, το αντικείμενο, αλλά και όταν υπάρχει ήδη ε, κάτοχος άδειας. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένας φορέας που είναι υπεύθυνος για τον υποέγκριση αντικείμενο. Και το τέταρτο είναι να διατηρηθεί η κατάσταση έχει και να μην προβλεφθεί ε, καμία καταβολή τέλους. Αυτές είναι οι τέσσερις εναλλακτικέ λύσεις. Πρέπει να διαβολευτούμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και υπάρχουν και πολλές άλλες εναλλακτικέ λύσεις που πρέπει να εξεταστούν ε, πριν ε, προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων. Όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως, η απουσία διαβαθμισμένων, ε, μάλλον κλιμακούμενων τελών, αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξεταστεί. Γνωρίζετε βέβαια ε, πόσο περίπλοκο είναι το θέμα των τροφίμων και τώρα ποικίλουν οι αιτήσει. Για να φέρω έτσι ενδεικτικά ένα πράγμα. Έχουμε γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, το σύστημα το γνωρίζετε όλοι σας, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες ε, εφαρμογές ε, όπως οι πρόσθετες ουσίες και άλλες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Το σύστημα στον τομέα των τροφίμων είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που ισχύει στον φαρμακευτικό τομέα, όπου ο οργανισμός φαρμάκων ε, έχει ε, σαφές αρμοδιότητες και ε, κανονισμούς από τη στιγμή που εγκριθεί ένα φάρμακο. Ένα πράγμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ο προϋπολογισμός. Οφείλουμε βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός της ΕΦΣΑ είναι σταθερός Δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουμε τον προπολογισμό, να τον αποδυναμώσουμε όταν θα συζητηθούν όλες οι εναλλακτικέ λύσεις. Όπως βλέπετε λοιπόν και κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της ε, μελέτης ε, της αξιολόγησης των επιπτώσεων υπάρχουν, ε, υπάρχει μια βεντάλια απόψεων και είναι πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς με σαφήνεια να αξιολογήσει το ύψος τελών για τους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα τρόφιμα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις, τις απόψεις όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων για να δούμε πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε λεπτομερέστερη αξιολόγηση επιπτώσεων ε, πριν καταθέσουμε τον κανονισμό, το σχέδιο κανονισμού. Ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε τη συζήτηση, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλα τέσσερα σημεία μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση. Σα προτείνω ή 20 λεπτά ένα ζήτημα να αφιερώσουμε. Άρα δίλεπτε, τρίλεπτε παρεμβάσει, όχι παραπάνω. Η 20 λεπτα ενα ζητημα να αφιερωσουμε αρα 3 λεπτές παρεμβασει οχι παραπανω η κυρια Ροτ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω η εκθέση είναι καλή. Εγώ ήμουνα πάντα ιδιαίτερα επιφλακτική όσον αφορά τα τέλη για την ΕΦΣΑ και αυτό για πολλούς λόγους. Διάβασα πολύ προσεκτικά τι αναφέρεται στην έκθεση για το θέμα της ε, ανεξαρτησίας και των τελών. Συμφωνώ με την ε, Κομισιόν, με αυτά που λέει. Αυτά που είπε ο εκπρόσωπος Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλά Ίσως το ότι η ΕΦΣΑ πρέπει ακόμα να διανύσει αρκετό δρόμο για να είναι σαφές ότι σε όλα τα θέματα η ΕΦΣΑ είναι ανεξάρτητη και ότι σε όλα τα θέματα γνωρίζει η ΕΦΣΑ ότι είναι σημαντική η αρχή της ε, πρόληψης. Στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου το ε, διαψώσαμε αυτό. Ε, η συνάδελφος Χαμογελάγια το ξέρει πολύ καλά η ΕΦΣΑ θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένη ως προς την πολιτική πραγματικότητα. Ε, αυτό ισχύει και για τους πρόεδρους των επιτροπών. Η κακή φήμη και η δυσαρέσκεια με τα αποτελέσματα που κατέθεσε η ΕΦΣΑ και η ε, κριτική απέναντι σε ανακοινώσεις του τύπου με οδήγησε στο να πω όχι, δεν επιθυμώ η ΕΦΣΑ ε, να βρεθεί σε σχέση με εισπραξη Αυτά που λέει η Κομισιόν στο έγγραφο είναι σωστά και συμφωνώ απόλυτα με την ε, περίληψη που αναφέρεται στη σελίδα 13 της έκθεσης και επίσης συμφωνώ και με αυτά που είπε ο συνάδελφος, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, σχετικά με τον κατάλογο ε, για τον οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, τέλη. Σωστό αυτό, να υπάρξει αξιολόγηση επιπτώσεων. Και όσον αφορά στις εναλλακτικέ λύσεις, εγώ πιστεύω ότι αν τελικά προχωρήσουμε σε σύστημα τελών, η εναλλακτική τρία είναι η καλύτερη. Και εκεί συμφωνώ με την Κομισιόν ως προς τα συμπεράσματά της και περιμένω να δω ποια θα είναι η μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και κυρίως ε, για το ότι περιμένατε τόσο πολύ να εξετάσετε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εγώ όμως ε, δεν καθόμουν στον καναπέ να καταβροχθίζω σοκολατάκια. Κάθε άλλο ε, από το πρωί είχαμε συζητήσεις για τον προπολογισμό που συνεχίζονται ακόμα. Είχα δουλειά λοιπόν και θέλω να επισημάνω ότι όλα τα τέλη τα οποία εμείς ε, καταβάλουμε ή μπορούμε να αποκτήσουμε για οποιοδήποτε οργανισμό, ε, τα τέλη αυτά προωθούν την ε, σταθερότητα μιας, ενός οργανισμού. Δεν προκαλείται αστάθεια, γιατί αν δούμε λιγάκι το τι κάνει ή το τι θέλει να κάνει το Συμβούλιο με τους διάφορους οργανισμούς δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί κάθε φορά να ορίσει τα όρια και να εγγυηθεί την σταθερότητα αυτών των οργανισμών. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτιμώ ε, να αποκτήσουμε αυτό που ισχύει ας πούμε για την ΕΜΕΑ, τον οργανισμό αυτό, για τον οργανισμό ΕΚΑ. Δηλαδή οι επιχειρήσεις ε, προσφέρονται στις υπηρεσίες και παρακαλώ πάρα πολύ οι επιχειρήσεις να καταβάλουν τα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και εγώ λοιπόν αυτήν την έκθεση τη βρίσκω ε, καλή. Ε, υπογραμμίζω, συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει το διαχωρισμό όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον και ε, τη δική μας την ευθύνη, τότε θα πρέπει να πληρώσει ε, ο Ευρωπαίος φορολογόμενος, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Εντάξει γι' αυτό. Όλα τα άλλα όμως όπου οι επιχειρήσεις ε, αν θέλετε κάνουν και διαφήμιση εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να εισαχθεί ένα σύστημα τελών. Πάρα πολύ καλό αυτό. Εγώ ελπίζω η Κομισιό να μην χρειαστεί άλλα πέντε χρόνια για να προβεί στην αξιολόγηση. Ελπίζω ότι δεν θα πρέπει να προβλέψουμε και πάλι αποθεματικό στον επόμενο προεπλογισμό για να αποκτήσουμε επιτέλους την πολυπόθητη αξιολόγηση. Ελπίζω η Κομισιόν να άκουσε περί τίνος πρόκειται και με το που θα βγει από την αίθουσα να τρέξει να δώσει την εντολή για αυτή την αξιολόγηση. Ευχαριστούμε κύριε Χόκ. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Θα ξανακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ μια παρατήρηση που απηχεί την παρέμβαση τη κυρία ε, Ντόκμαν ε, ε, Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τον προπολογισμό ενός οργανισμού. Λογικό αυτό. Απλώς ε, θα πρέπει να δούμε ότι η πρόταση φτάνει σε, ένα δύσκολο, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Τίθενται πολλαπλά ερωτήματα για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων και δεν πρέπει να ζητούνται τέλη Δηλαδή να ζητείτε ένα είδος παροχής υπηρεσιών που θα επιβαρύνει την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και στη συνέχεια όμως δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για τις επικείμενες γνωμοδοτήσεις. Ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα θέλατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων μου, παρακαλώ. Μάλιστα. Σε σχέση με την αξιολόγηση αντικτύπου θα πρέπει να πούμε ότι είναι μακρός τη διαδικασία, θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο, θα πρέπει να διαβουλευτούμε όλους τους εταίρους και να εξετάσουμε όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω το εξής. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τέλος για κάθε ένα από τα προϊόντα που καλύτερα να αξιολογήσει η ΕΑΤ. Δηλαδή, ε, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, πρόσθετες ουσίες, ε, συνήθως ουσίες ε, που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα ή για τις ζωοτροφές. Ε, ή ε, αιτιάσει ε, για την υγεία που καλύτερα να χειριστεί η Ευρωπαϊκή Αρχή ή τις διάφορες συμβουλές που ζητούνται από αυτήν την Ευρωπαϊκή Αρχή. Είναι πολλές και διαφορετικές αυτές οι λειτουργίες και άρα θα είναι εξαιρετικά δυσχερές για μας να προσδιορίσουμε το τέλος για κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες. Ε, πρέπει να αξιολογήσουμε τις ε, συνέπειες ε, αυτού του προσδιορισμού τελών και θα επανέλθουμε όταν έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη έκθεση μετά την έγκριση της αξιολόγησης αντικτύπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαγγέτε για τις διευκρινήσεις αυτές. Τώρα, σημείο 10 της Μεσίας Διατάξεως, επίσημη έλεγχη στα κράτη-μέλη για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών. Θα ακούσουμε ε, πρώτα τον κύριο Πουντλή. ο οποίος έχει συντάξει την έκθεση για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μας δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε την έκθεση που συντάξαμε. Ε, θα είμαι ταπεινόφρον διότι πρόκειται για την πρώτη έκθεση στον τομέα αυτό, ε, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 882 ε, 2002 για τους επίσημους ελέγχους ε, στα κράτη-μέλη. Είναι μια πρώτη έκθεση λοιπόν και θέλουμε να είμαστε μετριοπαθείς ως εκ τούτου. Το διαπιστώσατε κι εσείς ότι αποτελείται από τρία τμήματα η έκθεση. Πρώτα απ' όλα ε, παρουσιάζεται μία ε, σύνοψη των ελέγχων, ε, των δοκιμών, των εργαστηρίων των κρατών μελών. Κατόπιν, σε ένα δεύτερο τμήμα της η έκθεση εκθέτει τους ε, ελέγχους που έχει διεξαγάγει η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ ε, και η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ιατρικών Υπηρεσιών που κάνει τους ελέγχους στις τρίτες χώρες και τέλος πληροφορίες προέρχονται από άλλες πηγές που προέρχονται από την αγροβιομηχανία πληροφορίες που συλλέγουμε από τις μόνιμες επιτροπές της ε, πιστιστικής αλυσίδας ή πληροφορίες προέρχονται από το σύστημα ε, έγκαιρης προειδοποίησης που εμείς διαχειριζόμαστε από πλευρά της Επιτροπής. Ε, στα παραρτήματα της παραθέτει έκθεση 10 θεματικές υποεκθέσεις που παρουσιάζει ετησίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιρετικά διεξοδικές εκθέσεις. Ε, για τους ελέγχους για τις εγκεφαλοπάθειες, για τις ζωονόσους, ε, για τα, καταλή... Ε, για τα κατάλοιπα συγγνώμη, των παραστοκτώνων. Και... Έτσι γίνεται επισκόπηση των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί από τα κράτη-μέλη και η επιθυμία μας είναι να κάνουμε μία σχετικά σύντομη σύνοψη όλων των ελέγχων ε, που διεξήγαγαν τα κράτη-μέλη σε όλη την αλυσίδα, αρχίζοντας από τις ζωοτροφές, περνώντας από την ευημερία και την υγεία των ζώων, καθώς και τον έλεγχο της ασφάλειας της ε, τροφικής αλυσίδας. Ε, δυστυχώς, οι πληροφορίε που μας δίνουν τα κράτη-μέλη μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις που μας διαβιβάζουν, δύσκολα μπορούν να ε, αποτελέσουν αντικείμενο σύνοψης. Σε συνεργασία με την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικών Στοιχείων, σε στενή συνεργασία με την Eurostat και τα κράτη-μέλη, προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε συστήματα σύνταξη ηλεκτρονικών εκθέσεων ε, που εύκολα μπορούν ε, να μας οδηγήσουν σε ε, σύγκριση δεδομένων. Τώρα, προς το παρόν, προσπαθούμε να συγκρίνουμε μήλα με καρότα. Δύσκολα μπορούμε να βασιστούμε σε μη συγκρίσιμα δεδομένα. Γι' αυτό επανέρχομαι όπως είπα και στην αρχή, θα είμαστε μετριοπαθείς σε αυτή την έκθεση. Ε, ειλικρινά επιδέχεται βελτιώσεις και το γνωρίζουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε ε, μια πλούσια πηγή πληροφοριών για όλους τους εταίρου και για το Κοινοβούλιο, ε, κατά πρώτο λόγο, για τη βιομηχανία, για, τις, για τους καταναλωτές επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταδείξουμε ε, σε ποιο βαθμό ελέγχουμε την ε, διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Λίγοι λόγου χάρη γνωρίζουν πως τα κράτη-μέλη ε, διεξάγουν ελέγχους 8 εκατομμύρια δοκιμές για την τρελή αγελάδα για τις εγκεφαλοπάθειες ετησίως 80.000 περίπου δοκιμές για τα κατάλοιπα των παραστοκτόνων στην Ευρώπη. Λίγοι γνωρίζουν ότι πάνω από 600.000 ε, έλεγχοι γίνονται, ε, ε, βακτηριολογικοί έλεγχοι για τα τρόφιμα και θέλουμε να ενοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσουμε στις μελλοντικέ εκθέσεις. Αρχίσαμε ήδη να εργαζόμαστε θα εργαστούμε φυσικά αργά και για πολύ χρόνο διότι ε, πρέπει να ε, συνεννοηθούμε με όλες τις ε, συναρμόδιες εθνικές αρχές και να θεσπίσουμε ένα σύστημα βάσης δεδομένων και φυσικά τα κράτη-μέλη κατόπιν θα διεξαγάγουν τους ελέγχους και θα φτιάξουμε ένα ετήσιο συμπίλημα όλων των πληροφοριών. Τι σημαίνει αυτό, θα χρειαστούμε χρόνια για να τελειοποιηθούν οι εκθέσεις μέχρι ότου να είμαστε περήφανοι δηλαδή που, για την έκθεση που σας παρουσιάζουμε. Θα είναι μακρόχρονη διαδικασία οπωσδήποτε. Ε, γνωρίζουμε ότι δεν είναι τέλεια η έκθεση, ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ε, επικρίσεων. Ε, ξέρουμε ότι επιδέχεται βελτίωση και ε, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε. Ε, δεν έχουμε χρόνο, διακόπτη η Πρόεδρος. Όχι, όχι, παρακαλώ, έχετε ακόμη κάποια λεπτά αν ε, τα χρειάζεστε, γιατί κερδίσαμε λίγο χρόνο σε σχέση με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, γιατί μίλησε λιγότερο. Δεν έχουμε χρόνο αγόρευσης για τον εισηγητή, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα, οπότε έχετε περισσότερο χρόνο εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Τα, οι εκθέσει ε, των ε, κρατών μελών είναι σημαντική πηγή πληροφοριών για μας. Υπάρχουν ε, οι εκθέσεις ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κτηνιατρικού Οργανισμού και είτε μιλάμε για τα κράτη-μέλη είτε μιλάμε για τις τρίτες χώρες, δημοσιεύονται τα δεδομένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, προσβάσιμες πληροφορίες για όλους, ώστε να γνωρίζουν πώς έχει κατάσταση αναχώρα. Ε, ο στόχος μας εδώ δεν είναι να στιγματίσουμε το τάδι το δίνα κράτος μέλος ε, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καλύτερος και ο χειρότερος μαθητής, ε, ποιοι πρέπει να βελτιωθούν και ποιοι όχι. Δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος της έκθεσης. Πρόκειται για μεμονωμένες εκθέσεις ανά κράτος μέλος και καθής μπορεί να βρει εκεί τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αντίθετα, ο στόχος μας είναι μέσα στην έκθεση να καταδείξουμε το εξή και είναι σίγουρο ότι πρέπει να βελτιωθούν κάποια κράτη-μέλη, να καταδείξουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση για τη διατροφική αλυσίδα ανακράτος μέλος. Σας αρχίσω με τις ε, ήπιες, τις υπιότερες μεθόδους αν θέλετε. Υπάρχουν οι επιστολές, η ε, πίεση, οι εγκλήσεις, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να καλέσουμε το κράτος ε, να απευθύνουμε μια έκκληση στο κράτο μέλο ε, να κινηθεί αποτελεσματικότερα. Επίση, ρήτρε σε διασφάλιση, ώστε ένα κράτο μέλο ή μια τρίτη χώρα να επιβάλλει συγκεκριμένε ε, απαιτήσει ελέγχου για κάθε συγκεκριμένο προϊόν. Τέλος, ε, το ένα από τα πλέον αποτελεσματικά ή πλέον νομικώς ισχυρά μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η διαδικασία επί η διαδικασια επιπαραβαση ε, δεν ε, επιθυμούμε να κινήσουμε εμείς τέτοιες διαδικασίες διότι σήμερα Έχουμε περίπου 90 περιπτώσεις ε, τέτοιων διαδικασιών ε, επί παραβάση, 65 για τη μη μεταγραφή στην Εθνική Νομοθεσία των ε, Ενωσιακών Νομοθετημάτων και 24 για ουσιαστικές υποθέσεις. Τι εννοώ, μίζονες παραβάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, των φυτών, την ευημερία των ζώων ή την ασφάλεια των τροφίμων χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία, τα τεκμήρια, ε, με πυγμή ε, διότι πιστεύουμε προφανώς ότι όλα τα κράτη-μέλη, όποια και αν είναι αυτά και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και ουραγοί στην όλη διαδικασία, αλλά δεν θα κατονομάσω εδώ αυτά τα κράτη-μέλη, δεν θα τα στιγματίσω. Θέλουμε να μεριμνήσουμε ότως ώστε οι ουραγοί να βελτιωθούν ε, και να ε, φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό στάδιο ασφάλειας της διατροφικής αλυσίδας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το εξής. Η ε, η υπηρεσία τροφίμων και την ιατρική υπηρεσία κάνει περίπου 250 επιθεωρήσεις σε κράτη-μέλη και σε τρίτες χώρες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Περίπου το ίμιση ε, σχετίζεται με προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες ε, με ε, επισκέψει ε, πολυάριθμες επισκέψεις ε, ε, στις τρίτες χώρες αλλά και συνοριακούς ελέγχους κατά την εισαγωγή, δηλαδή επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη που φέρουν όμως επί ε, προϊόντων ε, φυτικών ζωικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. 50% των επισκέψεων που πραγματικά σχετίζονται με ε, επιθεωρήσεις κρατών μελών και 50% ε, αποστολών επισκέψεων στις τρίτες χώρες. Και προφανώς για τις τρίτες χώρες τα αποτελέσματα, τα πορίσματα των ελέγχων είναι προσβάσιμα για όλους. Ιδού, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ροτ έχει το λόγο. Όταν ε, ήρθα ερχόμενα στις Βρυξέλλες, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι σήμερα το απόγευμα θα ήταν όλο δικό μου ε, και όταν είδα την ημερήσια διάταξη ε, είδα με μεγάλη τα θέματα που ε, αναφέρονταν σε αυτή. Εγώ παλαιότερα ήμουν πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, για την ασθένεια των τρελών αγελάδων και σε όλα αυτά που προκύπτουν σήμερα να είναι η απόρρια αυτή της ε, παλαιότερης ιδιότητάς μου. Σήμερα ο ε, συνάδελφος ήταν ιδιαίτερα, επέδειξε ε, διπλωματική διπλωματικές ικανότητες. Εγώ όμως δεν θα το πράξω αυτό. Πρέπει να ομολογήσω ότι την έκθεση του FVO στην Ιρλανδία, την έκθεση αυτή δεν την είδα. Όμως θα επιθυμούσα στην έκθεση αυτή, στη δική μας, να αναφέρονται στοιχεία που να ευσταθούν. Χωρίς να χρειάζεται πάντα να παίζω το ρόλο του detective, θα έπρεπε να γνωρίζω, να μπορώ να γνωρίζω τι έκαναν τα κράτη-μέλη, πόσους ελέγχους, για ποιο λόγο και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ποιες είναι οι πληροφορίες που πήραν από τα κράτη-μέλη. Σέβομαι βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Πουντελέ, ότι δεν ε, θέλει να παίξει το παιχνίδι του name and shame, του να ονοματίζει τους... Ε, ε, Εγώ όμως θα ήθελα να το κάνω αυτό, να το κάνουμε. Είπαμε ότι έχουμε μια νομοθεσία ε, στα κράτη-μέλη για τα τρόφιμα που επιβάλλει αυτή η νομοθεσία το τι πρέπει να κάνουν, πόσους ελεγκτές να έχουν. Παρόλα αυτά όμως ε, τα κράτη-μέλη αμελούν αυτές τους τις υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν θέλω πια να είμαι τόσο συμπαθητική. Να δω. Ποια είναι τα ελλείμματα, σε ποιους τομείς υπάρχουν πραγματικές ελλείψεις. Μπορώ να το φανταστώ. Μπορώ μάλιστα να φανταστώ ακριβώς και την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν προβλήματα, αν θέλετε, και τις περιοχές και τα αντικείμενα. Όμως θέλω όλα αυτά να τα δω γραμμένα. Η έκθεση αυτή αναμφισβείται ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο, όμως αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής να είναι λίγο σαφέστερος στους αριθμούς. Ε, για τους συναδέλφους δεν ξέρουν πολλά για τους ελέγχους, ε, για τα τρόφιμα και ενδιαφέρονται, να τους πω ότι το έγγραφο είναι πολύ καλό για να το διαβάσουν. Εγώ ήξερα εκ των προτέρων πολλά, δεν ήξερα βέβαια τις λεπτομέρειες. Ίσως τώρα ο εισηγητής μπορεί να μου πει τώρα ποια, πόσοι έλεγχοι έγιναν, ποιε είναι οι εκθέσει των κρατών μελών, πόσα κρατημέλη δεν έδωσαν εκθέσει, ε, πόσα κρατημέλη ε, παρουσιάζουν δυσάρεστη εικόνα, πώς ε, εκπληρώνουν τα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους και ποιο είναι το αποτέλεσμα του οργανισμού FVO, Food and Veterinary Organization στην Ιρλανδία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέρεντ. Η κυρία Σεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κυρία Ροντμπέρεν, που είναι η συγγήτρια μας για τον κανονισμό, για τους ελέγχους, για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Γνωρίζω πολύ καλά τον κανονισμό και είναι σαφές ότι αυτή η έκθεση όπως είπε η κυρία Ροντ Μπέρεντ, ε, δεν είναι αρκετά πυκνή. Αλλά όπως είπε και ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να φταίει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με καρότα ε, και ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα. Μα είναι απαραίτητο αυτό για την ασφάλεια των τροφίμων, ούτως ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι με αποτελεσματικό τρόπο και να είμαστε σίγουροι ότι διεξαγάγονται με ομοιόμορφο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι έλεγχοι. Ε, εγώ είμαι στην Επιτροπή Γεωργίας και εκεί γίνεται μια σημαντική συζήτηση για τον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες. Και σε εκείνη τη συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παραγωγή τροφίμων και για τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας ε, και να το βελτιώσουμε όταν χρειάζεται. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε την σύνταξη εκθέσεων. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε ποια ζητήματα πρέπει να καλύπτουν οι εκθέσεις ένα άλλο σημείο το οποίο βλέπω με ιδιαίτερο σκεπτικισμό ε, και για το οποίο αγωνίστηκα πριν από 6-7 χρόνια είναι ο έλεγχος ε, της υγιεινής που γινόταν επί τη βάση κινδύνου. Επί το όταν επιστρέφουμε στην πραγματικότητα, Βλέπω ότι η αξιολόγηση κινδύνου είναι εξαιρετικά υποκειμενικό θέμα. Στη δική μου τη χώρα είδαμε ότι ε, στη, στα αγροκτήματα δεν σερβίρεται πια καφές και κουλουράκια γιατί δεν θεωρούνται ασφαλή. Ε, γιατί θεωρήθηκαν ε, μη ασφαλή αυτά τα κουλουράκια κανέλας. και στο σχετικό έγγραφα και στην έκθεση που συντάχθηκε διαβλέπουμε αυτούς τους κινδύνους και θα ήθελα ε, να πω το εξή, ε, ότι όταν εκπονήθηκε ο κανονισμό ε, για την ασφάλεια των τροφίμων στην περίοδο 2000 2004 επικράτησε πανικός στην Ευρώπη. πλήρη πανικός. Ήμασταν υπερβολικά τρομαγμένοι, μήπως υπερβάλαμε. Καλό θα ήταν να επανεξετάσουμε το θέμα των πρωτεϊνών, των ζωοτροφών. Υπάρχει έλλειψη ε, στην Ευρώπη και συνειδητοποιούμε ότι ε, πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να μην επικρατήσει ο κανιβαλισμός ε, στην Ευρώπη και να προσέξουμε τι κάνουμε με τις ζωοτροφές. Και το ίδιο ε, ε, ισχύει, προσοχή χρειάζεται για, για τις ε, κότες και για τους χείρους, δηλαδή θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα των πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές αυτών των ζώων. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζω και εγώ τα σχόλια των συναδέλφων. Θα βοηθούσε νομίζω να ακούσαμε, αν δεν θέλουμε να μιλήσουμε για κρατημέλη, μελη τέλος πάντων, κάπως να διευκρινιστεί για ποια προϊόντα πρόκειται και πού. Όσον αφορά τους ελέγχους, η ανησυχία δικιά μου είναι για την Ιρλανδία τουλάχιστον ότι είχαμε ε, με διοξίνες ε, μόλυνση τροφίμων και χρειάζεται και αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου, αλλά και δράση. Δεν ξέρω σε τι βαθμό η έλεγχη μας είναι απλώς στα χαρτιά και δεν πρόκειται για πραγματικούς ελέγχους με προβλήματα που υπάρχουν στην υγιεινή, την ασφάλεια κλπ. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια της κυρίας Πόλσεν για τρίτες χώρες και τους ελέγχους εκεί, Έχουμε το ίδιο επίπεδο επιθεωρήσεων και ελέγχων στα τρόφιμα που ελέγχουμε όπως και στα, ε, που εισάγουμε, συγγνώμη, όπως και στα τρόφιμα που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Και κυρίως, όπως είπα και πριν, πού υπάρχουν, σε ποιες περιοχές υπάρχουν τα προβλήματα κυρίως. Ευχαριστούμε. Κύριε Κλάς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και το θέμα αυτό ε, δεν μπορεί κανείς ε, να το ε, εξετάσει με αυτούς τους πολύ ε, γυμνούς αριθμούς. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεωρώ ότι εξαντλείται το έργο μας με το να συγκεντρώνουμε στοιχεία. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση περιεχομένου. Όσον αφορά λοιπόν σε αυτή την αξιολόγηση που εγώ τη θεωρώ αυτονόητη, επ' αυτής ε, θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να μας πει η Κομισιόν πώς μπορεί να διασφαλίσει ότι στην περίπτωση που εφαρμόζεται το πακέτο υγιεινής ότι πράγματι θα εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή αφενός προβλέπεται κάποια ευελιξία, όμως και οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται τη νομική ασφάλεια. Εγώ λοιπόν μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν ε, θεωρώ ότι πρέπει να πούμε και κάτι <coughs> επί της ουσίας. Και ε, το ερώτημα είναι ποια ακριβώς νομική ασφάλεια μπορεί να προσφερθεί στις αρμόδιες αρχές επιτόπου. Ποιος άλλος θέλει το λόγο? Κρήτον. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες και χρειαζόμαστε επίσης και στοιχεία για, τους, για τις συνέπειες των ελέγχων. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι που μας πέρασε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, διαπιστώσαμε ότι παράνομα η πατάτα, η γενετικά τροποποιημένη καλλιεργιόταν φυσικά φταίει το κράτος μέλος, φταίει η επιχείρηση η οποία πούλησε τους σπόρους. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποιες είναι οι συνέπειες των ελέγχων. Il θέλει το λόγο παρακαλώ. Ποιο θέλει το λόγο άλλος. Όχι, λοιπόν, για να μα πείτε λοιπόν εσείς τη Κομισιόν, για προσπαθήστε να μα φωτίσετε λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία Ροτ Μπέρετ πρώτα. Για το πόσε χώρε απάντησαν. Μία δεν απάντησε την πρώτη αυτή αξιολόγηση του 2007. Μία. Αλλά είναι πολύ. Δεν έπρεπε. Το 2008 φροντίσαμε να έχουμε απαντήσεις από όλες τις χώρες. 2007 ήταν η πρώτη φορά που προβήκαμε στον χείρημα αυτό. Και το ξέρουμε, δεν είναι τέλεια η κατάσταση, θέλουμε να τη βελτιώσουμε. Θέλω να απαντήσω τώρα και στην κυρία Πόλσεν. Θέλω να διευκρινίσω ένα σημείο το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Είναι το θέμα αυτό των γλυκών που φτιάχνουμε στο σπίτι και τα πουλάμε για να μζέψουμε λεφτά για να τα δώσουμε στους στοχούς ας πούμε. Ε, λοιπόν, ποτέ δεν έχει διακανονιστεί από κοινωτική άποψη αυτό το πρόβλημα. Έχει βγει επίτηδες από το κεφάλαιο υγιεινής και είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες το διακανονίζουν. Συνεπώς δεν θα απαντήσω εγώ αν είναι καλό ή κακό, που οι γιαγιάδες ή τέλος πάντων οι γυναίκες φτιάχνουν γλυκά και τα πάνε μετά στην εκκλησία και τα πουλάνε για να μαζέψουν λεφτά. Οι άντρες, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, και οι άντρες. Εντάξει, πιο σπάνια, αλλά ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, ναι. Εδώ κάνω μια διάκριση φιλεκτικού χαρακτήρα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Είναι λοιπόν κάτι που το κανονίζουμε σε εθνικό επίπεδο. Επίτηδε το αφήσαμε απ' έξω, γιατί σκεφτήκαμε ότι οι εθνικές αρχές, οι περιφερειακές, οι τοπικές μπορούν πολύ καλύτερα να κανονίσουν αυτό το θέμα. Και εμείς έτσι καλώ να σας πω την αλήθεια, είμαστε υπέρ. Πρέπει να βοηθάμε τις εκκλησίες, όποιο δόγματος και αν είναι αυτές. Τώρα, για τα κρεατάλευρα τώρα, το 2011 θα έχουμε ένα σχέδιο και ο κανιβαλισμός, κανιβαλισμός. Μπορείτε λοιπόν να επαληθεύσετε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς δεν σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε τον ε, κανιβαλισμό σε τέτοιου είδου μελλοντικέ αδειοδοτήσει. Το θέμα τώρα τη διοξίνη ε, στο χείριο κρέα ε, στην Ιρλανδία. Μα ακριβώ επειδή υπήρχαν ελέγχοι σε αυτό το κρέα, γι' αυτό ακριβώ βρέθηκε και η κακή χρήση, πώς δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν μολυσμένα έλαια και βρέθηκε το πρόβλημα. Ακριβώ επειδή υπάρχουν έλεγχοι. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν το βρίσκουμε. Και το χείριο κρέα θα εξακολουθούσε να έχει διοξίνη και να το τρώγαμε. Ακριβώ όμω επειδή υπάρχουν έλεγχοι, η Ιρλανδική κυβέρνηση με εμά, αλλά η Ιρλανδική κυβέρνηση πήρε πολύ αυστηρά μέτρα. Έξι μήνες παραγωγής χείριου κρέατος αποσύρθηκαν από την αγορά. Χάρη στους ελέγχους αυτούς επαναλαμβάνω. για, την, ε, για τα γιόμιλα, τα γενετικά τροποποιημένα. Μόλις το μάθαμε, αμέσως ήρθαμε σε επαφή με την ε, σχετική επιχείρηση για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Αν υπήρχαν ε, γιόμιλα που είχαν εμολυνθεί από μη επιτρεπόμενα γιόμιλα γενετικά τροποποιημένα, θα έπρεπε να καταστραφούν. Η επιχείρηση όμως καταστρέφει 200 με 250 τόνους γεωμήλων, 200 με 250 τόνους, κυρίως από τη Σουηδία και θα καταστραφούν πλήρως και δεν θα πάνε στη βιομηχανία. Ξέρετε ότι τα γεώμηλα αυτά, τα γενετικά τροποποιημένα, δεν είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Πάνε στη βιομηχανία για να φτιάχνετε άμυλο για, χάρτη, για χαρτί. Ποτέ δεν ε, φτάνει στην ανθρώπινη κατανάλωση. Τα γιόμιλα αυτά λοιπόν που μολύνθηκαν σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. 0,01% θα καταστραφούν όλα. Δεν θα μπουν σε καμιά αλυσίδα ούτε βιομηχανική ούτε διατροφής, ούτε για ζωοτροφές. Θα το προσέξουμε πάρα πολύ σοβαρά με πλήρη συνεργασία με τις Σουηδικές Αρχές που βρίσκονται επιτόπου. τόπου. Τέλος, τέλος, πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στις τρίτες χώρες. Πρέπει να σας πω ότι τα προϊόντα τρίτων χωρών, είτε επειδή δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις επί τόπου, στις χώρες δηλαδή από τις οποίες εισάγουμε τρόφιμα, εμείς επικεντρωνόμαστε πολύ περισσότερα, περισσότερο στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, είτε πρόκειται για λακτοκομικά, για μέλι, για κρέας, ψάρια. Εκεί υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι και για την ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για ζωοτροφές. Είναι λοιπόν επικίνδυνα φέρουμε εμείς προϊόντα και γι' αυτό κάνουμε επιθεωρήσεις πολύ περισσότερο σε αυτά τα προϊόντα στις τρίτες χώρες, παρά σε άλλα προϊόντα όπως είναι η ζάχαρη. Για παράδειγμα, και ξέρετε ότι εισάγουμε πολύ ζάχαρη από τρίτες χώρες. Επαληθεύουμε λοιπόν με τις επιτόπου επιθορήσεις που κάνουμε ή με ελέγχους ε, που γίνονται στα σύνορα ότι τηρούνται οι κοινοτικοί κανόνες. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν τελικά στις αγορές μας είναι προϊόντα τα οποία είναι εντελώς αντίστοιχα υγειονομικά με τα ε, δικά μας ευρωπαϊκά προϊόντα. Στα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τις τροφές και τις ζωοτροφές, στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βλέπετε ότι οι περισσότερες έχουν να κάνουν με προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ελέγχουν το τι γίνεται στις τρίτες χώρες και τα προϊόντα αυτά και αν δεν είναι κατάλληλα επιστρέφονται στην χώρα προέλευσης ή πάνε σε άλλες τρίτες χώρες που δυστυχώς δεν κάνουν τόσους ελέγχους όπως εμείς. Θα ετοιμάσουμε μια έκθεση για τα τέλη του 2010 για όλους αυτούς τους ελέγχους που κάνουμε όσον αφορά την εισαγωγή τροφίμων από τρίτες χώρες όπως επίσης και για την εισαγωγή ζώων και φυτών. Επί τη ευκαιρία αυτή θα συζητήσουμε μαζί σας και με άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε, να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε τους ελέγχους στις τρίτες χώρες. Ακόμα σήμερα υπάρχουν τομείς που ελέγχονται πολύ λιγότερο, εναρμονίζονται λιγότερο. Υπάρχουν τομείς στους οποίους ελοχεύουν λιγότεροι κίνδυνοι. Όμως θα εκπονήσουμε μία μελέτη για το προϊόν, το κίνδυνο και το, τη χώρα προέλευσης, για το τρίγωνο αυτό, ώστε να φτιάξουμε ένα προφίλ κινδύνου και να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα σύνορα. Κίνδυνος και προϊόν είναι ένα δίδυμο το οποίο αξιολογείται από την υπηρεσία μας. Και ο παράγοντας χώρα προέλευσης είναι ένα κριτήριο πολιτικό όχι επιστημονικό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που όσον αφορά τον έλεγχο των τροφίμων βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με εμά. Άλλες όχι, δυστυχώς. Αυτά λοιπόν για να σας πω ότι στα τέλη της χρονιάς και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν την έκθεση αυτή για τους ελέγχους των ε, τροφίμων, ζώων και φυτών. Ευχαριστούμε κύριε Μπουτλέ. Τώρα περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισητιστικής ασφάλειας. Έχουμε τον κύριο Μπερλάτο η συγητή για τις γνωμοδότησής μας. Κύριε Μπερλάτο, θέλετε να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ε, η πρώτη, είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί ασθένειες ε, όπως οι τρελές αγελάδες, τα σκάνδαλα σχετικά με την παραποίηση προϊόντων και τικετών, όλα αυτά ευαισθητοποίησαν τους καταλωτές που ζητούν καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και πρέπει να αναφέρουμε ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται έχοντας κατά νου ότι οι προβλέψεις λένε ε, θα έχουμε μέχρι το 2050 αύξηση κατά 40% του πληθυσμού, άρα δηλαδή μέχρι τότε θα υπάρχει και πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης τροφίμων. Νομίζω ότι ε, πρέπει να δώσουμε τις ε, απαραίτητες απαντήσεις και σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν αλλά και στους άλλους. Όσοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν, ε, αυτοί ε, θέλουν όλο και πιο ποιοτικά προϊόντα. Η δυνατότητα επιλογής Ισχύει για μερικούς αλλά και για άλλους, όπως σας είπαμε δεν ισχύει. Αρκετοί είναι αναγκασμένοι ε, να κάνουν οικονομία ακόμα και εις βάρος της ε, υγείας τους. Υπάρχει μια, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων, όμως ε, και σε αυτούς πρέπει να εγγυηθούμε ένα ελάχιστο κατώτατο όριο επισητιστικής ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων. Η επισητιστική ασφάλεια και ε, το δικαίωμα σε αυτήν, αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε μέσα από τη σωστή ενημέρωση και την ε, ετικετοθεσία. Η γεωργική δραστηριότητα με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ε, διδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι καλλιεργητές δεν ασχολούνται με ε, τις καλλιέργειες ε, γιατί τους αρέσει αλλά γιατί το έχουν ανάγκη. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και η προστασία αυτού έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα των προϊόντων άρα και για την επιστημιστική ασφάλεια. Η οικονομική κρίση ε, που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να επενδύσει στη γεωργία και στον τομέα των τροφίμων και μέσα από συχνούς ελέγχους ε, οι οποίοι θα διαπιστώνουν κατά πόσον εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Η ε, πρόταση γνωμοδότησης που κατατίθεται είναι ανοιχτή και με μεγάλη μου χαρά θα δεχθώ ε, συμπληρωματικές παρατηρήσεις εκ μέρου των συναντέλφων και βεβαίω με μεγάλη μου χαρά θα προσπαθήσω να τι εξετάσω και να τι χρησιμοποιήσω για να βελτιώσω την πρόταση που έχω καταθέσει. Ωραία. Θα ξεκινήσω από τους σκιώδη εισηγητές. Ο κύριο Κύριλοφ πρώτα. Sì, io sono italiano, l'ho detto in aula l'altro ε, εγώ λέγομαι Πυρίλο, Ιταλός είμαι. Το Πυρίλιο είναι στα Ισπανικά, Πυρίλο, χωρίς G. Εντάξει, ε, ίσως ε, με συγχωρείτε που το είπα, αλλά ήθελα να το διευκρινίσω. Την άλλη φορά ε, ίσως η πρόεδρος θα ε, καταφέρει να προφέρει σωστά το όνομά μου. Θα προσπαθήσω, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Περλάτο για την έκθεσή του, διότι η έκθεση αυτή καθιστά, προβάλλει ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για την ψηφιστική ασφάλεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια που σχετίζονται και με τη γεωργία, όχι μόνο την ευρωπαϊκή αλλά την παγκόσμια. Προκλήσεις ε, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς μόνο εφόσον σκεφτούμε ότι είναι συμπληρωματικές ε, οι προκλήσεις ε, που υπάρχουν αν λάβουμε υπόψη στις επόμενες δεκαετίες θα αυξηθεί η ζήτηση για τρόφιμα, αυτό σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητο να καλυφθεί η ζήτηση αυτή και βεβαίως αυτό ε, συνεπάγει ότι θα πρέπει όλα αυτά να συμβαδίζουν με την ασφάλεια. Η ΦΑΟ, ο οργανισμός, ο παγκόσμιος προβλέπει ότι θα περάσουμε στα 9 δις ε, κατοίκους ανά τον κόσμο μέχρι το 2050 και ως εκ τούτου ε, η αύξηση αυτή θα ε, επηρεάσει κυρίως τις αναδιόμενες οικονομίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετείται και αυτό στα θέματα ψεπιστικής ασφάλειας. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τροφή ασφαλής και θρεπτική. Αυτές θα πρέπει να είναι οι αρχές που θα ε, καθορίζουν τη στάση της Ευρώπης ε, στις προτάσεις που θα καταθέσει. Ε, όμως ε, μπορεί αυτό να το πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν αν δεν υπάρξει επέμβαση στις ασύμετρες νομοθετικές δυνάμεις που εξακολουθούν να υπάρχουν και αφορούν στην παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή λοιπόν υπάρχει παγκοσμιοποίηση των αγορών και προφανώς ε, τα τρόφιμα ε, εμπίπτουν σε αυτή την παγκοσμιοποίηση, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ε, στην ευσυντητική ασφάλεια, όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και σε αυτά ε, που καταναλώνονται στην παραγωγή αλλά και στην κατανάλωση. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόζει μεγαλύτερη αυστηρότητα την αρχή της αμοιβαιότητας ε, των κανονισμών. Να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει για την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, στις συζητήσεις που γίνονται για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, δεν αρκεί να λέμε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να ενισχύσει την ψηστική ασφάλεια. Να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να ενισχύσει και την ασφάλεια των προϊόντων που καταναλώνονται στην Ευρώπη. Η παγκοσμιοποίηση βέβαια απαιτεί να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίες επηρεάζουν τα μάλα, τις τιμές και έχουν πάρα πολλές συνέπειες ακόμα και στην επισητιστική ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση που γίνεται για θέματα ασφάλειας ε, ε, φοδιασμού με τρόφιμα δεν μπορεί να αποκρύπτει και τις επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν για το περιβάλλον οι βιολογικές καλλιέργειες είναι όλο και πιο απαραίτητες. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σκαλλιέργειες αυτές ακόμα και έξω ευρωπαϊκές χώρες. Για το θέμα του περιβάλλοντος, εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουν οι έρευνες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ε, ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική βοήθεια από την χρήση της βιοτεχνολογίας. Γιατί εδώ μιλάμε για τεχνικές που όχι μόνο επιτρέπουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια στον εφοδιασμό, παράλληλα επιτρέπουν και να αποβάλουμε τα ζυζάνια τα οποία πλήττουν τις βιολογικές καλλιέργειες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πυρίλο. Καλό. Ο κύριος Ουγιάς παρακαλώ τώρα. Merci. Grazie Corinne. Eh, la mia eh, valutazione sul parere che η δική μου η αξιολόγηση για αυτά που μας είπε ο κύριος Περλάτο, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το ότι αυτό που είπε στο τέλος, ότι είναι ανοιχτός, είναι μια γνώμη ανοιχτή και νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε για να ενισχύσουμε λιγάκι, να εμπλουτίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση, όπως το έκανε τώρα ο ε, κύριος Πυρίλο. Αν δούμε το θέμα κάτω από αυτό το πρίσμα, τότε θέλω να σας πω ότι οι φιλελεύθεροι προτείνουν μέσω εμού ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί κυρίως και το θέμα της γεωργίας. Βεβαίως δεν εμβαθύνουμε σε περιβαλλοντικά θέματα τα οποία αφορούν αυτήν την Επιτροπή. Ως εκ τούτου πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε να έχουμε μια γεωργία ε, συμβατή με το περιβάλλον, μια γεωργία που θα επιτρέπει να προωθηθούν ε, τα περιβαλλοντικά θέματα για να αποκτάμε ποιοτικά και υγιή προϊόντα. Πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει ε, παραγωγικότητα και προστασία περιβάλλοντος. Να κατανοήσουμε αυτά τα δύο θέματα πάνε μαζί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι λάθος το ότι στη γνωμοδότηση δεν γίνεται καμία αναφορά στην κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να ε, προσθέσουμε αυτό ε, το οποίο πρέπει να ενταχθεί στη μεταρρύθμιση της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Κατά την άποψή μας, όπως επίσης πιστεύω ότι στη γνωμοδότηση ε, πρέπει να γίνεται και αναφορά στα αυτά που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, ο ΦΑΟ. Να πω και κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην παράγραφο 2 θα πρέπει η παράγραφος αυτή να γίνει πιο ισχυρή ε, μια τροπολογία που να κάνει αναφορά στην τρέχουσα οικονομική κρίση, στην κρίση του τομέα, στην Ευρώπη και σε διάφορα άλλα μέρη. Όσον αφορά στην παράγραφο 3, νομίζω εκεί πρέπει να αναφέρουμε ότι μόλις πριν από λίγο εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο δύο εκθέσεις. Εκθέσεις που αφορούν στην σύναψη ε, συμφωνιών ε, με ε, τους μεγάλους διανομής. Νομίζω ότι είχαμε την έκθεση Μπουβέ επ' αυτού του θέματος. Άρα δηλαδή μπορούμε να επαναφέρουμε τέτοιου είδους επιχειρήματα, όπως επαναφέραμε και την έρευνα για τους μεγάλους διανομής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε επικοδομητική στάση απέναντι στην γνωμοδότηση, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί και να πούμε ότι αυτά που ε, περιγράφει η παράγραφος 7 σχετικά με την ασφάλεια είναι σημαντικά. Τέλος, να πω ότι καταλαβαίνω βέβαια ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του προσέγγιση, αλλά κατά δική μου άποψη, μια τροπολογία για το ρόλο των ε, μεταλλαγμένων προϊόντων, ε, μια τέτοια τροπολογία πρέπει να την καταθέσουμε. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε όλοι, αλλά τελικά ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταθέσουμε μια τροπολογία για τα μεταλλαγμένα προϊόντα σε αυτήν την έκθεση. Φερέρα. Αλλά τρία λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω κύριε Φερέρα. Ναι, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση ε, του εισηγητή. Ε, σημειώνουμε πρόοδο για σημαντικά σημεία, όπως ε, ε είπαν και οι συνάδελφοι και πρόσθεσαν και άλλα σημεία που πρέπει να πραγματευτούμε εδώ. Δεν έχουμε χρόνο, οπότε θα αναφερθώ στα δύο-τρία ε, σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου στοιχεία. Πρώτον, η επιστημιστική ασφάλεια και η οικονομική κρίση. Το θέμα της μεταβλητότητας των τιμών ε, υπάρχει η δυνατότητα κερδοσκοπίας για τις τιμές των τροφίμων. Πρέπει να το παρεμποδίσουμε αυτό. Πρέπει να παρεμποδίσουμε αυτή την κερδοσκοπία γιατί έχει τραγικές επιπτώσεις ως προς τη μεταβλητότητα των τιμών. Διάφορες υποσχέσεις ε, σε σχέση με την κατάργηση κάποιων ε, ε, παραγόγων και χρηματοπιστωτικών μέσων που επιτρέπουν την κερδοσκοπία δεν έχουν υλοποιηθεί. Μιλώ για παράγωγα παραδείγματος χάρη που επιτρέπουν ε, αυτή την κερδοσκοπία για τα τρόφιμα ε, και που μας οδηγούν ε, σε εκρηκτικές καταστάσεις από κοινωνικής πλευράς όπως είδαμε στη Μοζαμβίκη παραδείγματος χάρη πριν από λίγες εβδομάδες τέλος πρέπει να διακόψουμε την κερδοσκοπία να σταματήσουμε την κερδοσκοπία Αυτά για την, ε, το συνδυασμό της εμπορικής πολιτικής και της επιστημιστικής ασφάλειας. Επίσης, ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και η εξασφάλιση του. Ε, τι απαιτεί, ε, να α, επαναπροσανατολιστεί το διεθνές εμπόριο, να ακολουθήσει τη λογική της συμπληρωματικότητας και όχι τη λογική του ανταγωνισμού ανάμεσα στη, στους παραγωγούς και τις παραγωγές. νομίζω ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να το καλύψουμε μέσα στην έκθεση. Ένα άλλο θέμα θέμα τώρα είναι η κοινή ε, γεωρική πολιτική που αναφέρθηκε και θα πρέπει να τύχει διεξοδικότερης ανάλυσης ε, μέσα στην έκθεση. Είναι κατεπήγον πρέπει να παρεμποδίσουμε αυτήν την μείωση της βιοπικιλότητας ε, των ζωικών και φυτικών ειδών που συνδέονται με την διατροφή των ανθρώπων. Δηλαδή σήμερα αυτό αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα και πρέπει να το χειριστούμε οι ισχύουσε πολιτικέ και συγκεκριμένα η κοινή γεωρική πολιτική συμβάλλει στην φθήνουσα ε, βιοπικιλότητα ε, την ε, μειωμένη ποικιλότητα των ζωικών και φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση. Πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε αυτό το θέμα για την προστασία των περιφερειακών ποικιλιών των συγκεκριμένων παραγωγών, ε, δηλαδή της παραγωγής συγκεκριμένων περιοχών και ε, αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιμένους περιοχές. Ε, Τέλος, η επισητιστική ασφάλεια έχει άμεση σχέση με την επισητιστική κυριαρχία. η κυριαρχία των κρατών μελών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δηλαδή, ε, ξέρετε, υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σοβαρά ελλείμματα στον ισολογισμό ε, τον επισητιστικό του ισολογισμό και πρέπει για να κατοχυρώσουμε την επισητιστική ασφάλεια. Ναι, ναι, τελειώνω, Πρόεδρε. Πρέπει λοιπόν ε, ε, τα εντατικά μοντέλα να καταργηθούν και διακόπτει η Πρόεδρος. Ε, τέσσερις. έχουν ζητήσει ακόμα το λόγο, αλλά να είστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το τελευταίο θέμα. Τάκμαρ Μπέρεν είναι η πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω εκ μέρους Τασιάν Σάμου, που είναι η συγκήτρια. Ήταν εδώ όλο το απόγευμα, αλλά έπρεπε να φύγει να πάει στο αεροδρόμιο. Ζητά συγγνώμη και εκ μέρου τη λοιπόν σα λέω ότι χαιρόμαστε για την έκθεση αυτή του κ. Παγάτη. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται να δούμε το πράγμα της αντιστάθμισης των απολειών και το θέμα της επιζητιστικής ασφάλειας. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες, μου είπε ότι βρίσκει, που θέλει να υποστηρίξει. Ιδιαίτερα τονίζει η κυρία Τεσιάνα Κτάβια Σαρμπού ότι και στην ε, Επιτροπή Γεωργίας θα φροντίσει να τονίσει το θέμα της χρήσης γης, της διαθέσιμης γης και θα φροντίσει το ΣΥΠΗ να δεχτεί αυτό το μέτρο. Η οικονομική στήριξη τώρα για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα πρέπει να μην ε, καταστρέφει, μάλλον να συνάδει με την ζήτηση των τροφίμων και τις ανάγκες που υπάρχουν για τρόφιμα. Η εξάρτησή μας πρέπει να μειωθεί. Μου ζήτησε επίσης να σας πω ότι πρέπει να δούμε την βιολογική γεωργία. Διότι είναι πολλά το φέλη από τα βιολογικά προϊόντα στον κύκλο της φύσης. Τέλος. Αυτά είναι τα κύρια νομίζω και για μια φορά συγγνώμη. Θα επανέλθει βέβαια κάποια άλλη φορά σίγουρα θα υποβάλει και τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σνάλφο Μπερλάτο, ο οποίος υπέβαλε μια θαυμάσια έκθεση και κυρίως ε, κατάφερε ε, όλες απόψεις να τις συμπεριλάβει σε μία και μόνο σελίδα. Θέλω να υπενθυμίσω στους ε, συναδέλφους ότι εδώ συντάσσουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γεωργίας και δεν χρειάζεται να επανανακαλύψουμε τον τροχό. Έχουμε, θα έχουμε να κάνουμε με εκατοντάδες τροπολογιών και δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την, ή να εντάξουμε τις παρατηρήσεις μας στην Επιτροπή ε, που θα γίνει στην Επιτροπή Γεωργίας. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει τις ευθύνες της, αυτό είναι σαφές και προβάλλεται και εδώ θέλω να μιλήσω για την ολοκληρωμένη γεωργία και να προσθέσουμε αυτή τη λέξη. Δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση όπου θα ήθελα να παρακαλέσω την προσοχή του κ. Μπερλάτο. Στο σημείο υπαριθμών οποία αναφέρεται ότι τα ε, τρόφιμα θα πρέπει να είναι προσιτά για τους ε, καταναλωτές. Και εδώ νομίζω άνετα μπορούμε και να προσθέσουμε ότι και οι παραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν τις ε, σωστές τιμές για τα προϊόντα τους. Αυτό ταιριάζει πολύ καλά. Έγινε ήδη λόγος από τους άλλους ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα εποχικά και στα περιφερειακά προϊόντα. Αυτό ε, πρέπει να το ε, πούμε στην κοινωνία μέσα από την ενημέρωση και από την καλή και ε, αν γίνουν τελικά όλα αυτά νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να στηρίξω, λέει ο κύριο τα σχόλια της Δασιάνα Σαρβού. Ακούστηκε στην αίθουσα αυτή η κερδοσκοπία αυτή την εποχή στις τιμές. Είναι γνωστό ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντί να ασχολούνται με τον Άστακ, άρχισαν να ασχολούνται <coughs> με το δημόσιο χρέος των χωρών και με τις τιμές των τροφίμων. Γι' αυτό και το 2008 είχαμε, παρόλο που είχαμε τη μεγαλύτερη παραγωγή είχαμε στα Δημητριακά, είχαμε την μεγαλύτερη κρίση ποτέ στα Δημητριακά, αν είναι δυνατόν. Ένα άλλο θέμα <coughs> είναι η απώλεια δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πάνω στους πόρους. Ισχύει για την Ινδία, είναι γνωστό. Ξέρουμε τι καταστροφή επέφεραν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στην Ινδία, όπου εκεί οι ακρότες είχαν σπόρους που ήταν προσαρμοσμένοι στο τοπικό περιβάλλον και μπορούσαν να τους ε, χρησιμοποιούν. Μετά τους είπανε ότι οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι θα ήταν προτιμότεροι. Γιατί δεν θα χρειαζόντουσαν παστοκτόνα κτλ. Οπότε μετά έπρεπε να πληρώνουν αυτούς τους σπόρους. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε την ελεύθερη πρόσβαση στους σπόρους. Πρέπει να μπορεί ακόμα και δεν έχεις χρήματα να καλλιεργείς κάτι. Γιατί αλλιώς θα έχουμε ξανά κρίση τιμών στα τρόφιμα. Ο κύριος Νίκολσον τώρα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση. Άκουσα τη συζήτηση και σήμερα το πρωί. Η ασφάλεια τροφίμων είναι ένα πράγμα που δεν μπορείς να εγγυθεί στο σημερινό κόσμο όσο και προσπαθήσεις. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να υπάρχει προμήθεια στο μέλλον. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να μπερδεύουμε την ε, ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά την προμήθεια με, την, ε, με τα ασφαλή τρόφιμα. Το άλλο θέμα είναι οι αλλαγές στις τιμές. Ούτε και αυτό είναι εύκολο. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλει κανείς να έχει εφοδιασμό τροφίμων σε καλές τιμές, λογικές, για όλους, τότε πρέπει να μελετηθεί εκ των προτέρων η παραγωγή. Ποτέ όμω δεν μπορεί να λάβει υπόψη σου τα πάντα, τι θεομηνίε, για παράδειγμα πλημμύρε, ξηρασία, δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί ο νομοθέτη να τα προβλέψει αυτά και να κάνει κάτι για αυτά. Άρα, για να έχουμε ασφαλή εφοδιασμό, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιε αβεβαιότητε. Τα ψηλέ τιμέ, χαμηλέ τιμέ. Αν έχει χαμηλέ τιμέ, ε, η παραγωγή δεν ε, παράγουν αρκετά και πρέπει να εισάγουμε τρόφιμα που παράγονται με προδιαγραφές άγνωστες σε μας, με ελέγχους άγνωστους σε ενώ εκεί μπαίνει το θέμα ε, του ασφαλούς τροφίμου. Μην ε, υπερρυθμίζουμε τις αγορές μας γιατί αυτός είναι ένας κίνδυνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά, για να ολοκληρώσουμε δύο λόγια. Δεν έχουμε χρόνο, λυπάμαι. Έχουμε πέντε λεφτά στη διάθεσή μα για το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, κυρία Μαγκίνε. Ναι, αλλά τότε τι θα γίνει με το επόμενο. Εντάξει, ναι, αν θέλετε, εντάξει. 30 δευτερόλεπτα. Πολύ σύντομα. Πρέπει να υπογραμμίσω το εξή θέμα μπερδεύουμε τον ασφαλή εφοδιασμό με τα ασφαλή τρόφιμα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να υπάρχει μπέρδεμα και στη μετάφραση, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο έννοιες. Αν μας απασχολεί η βιοπικιλότητα που χάνεται, πρέπει να διατηρήσουμε τους οικοτόπους που παραμένουν και η εντατικοποίηση της γεωργίας κινδυνεύει να καταστρέψει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε βιώσιμη γεωργία. Αυτή είναι στην καρδιά της πολιτικής μας και πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στην έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν κύριε Σιγητά, ευχαριστώ για την τόσο καλή σας έκθεση. Θέλω να ε, τους συναντέλφους ότι θα συμπεριλάβω τις ε, προτάσεις τους ε, για να βελτιώσω τη γνωμοδότηση. Και θέλω και να τους ενημερώσω ότι και εγώ ίδιο μπήκα στον ε, πειρασμό να γράψω πολλά περισσότερα, αλλά τελικά έπρεπε να αντιμετωπίσω και να καλύψω δύο ανάγκες. Πρώτον, η γνωμοδότηση να παραμείνει μέσα ε, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γιατί επί της ουσίας είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Γεωργίας. Και από την άλλη, ένα θέμα που έπρεπε να καλύψω ήταν ότι έπρεπε να είμαι ε, περιορισμένος και περιεκτικός. Ε, αυτή ήταν η εντολή και η σύσταση που είχα. Βεβαίως, εφόσον κατατίθενται τροπολογίες, με μεγάλη μου χαρά να λάβω υπόψη μου τις προτάσεις ε, και ευχαριστώ όλους εκείνους που διάβασαν προσεκτικά την πρότασή μου. Και ε, προφανώς λείπουν αρκετά πράγματα διότι όπως σας είπα είτε διότι έκρινα ότι δεν ήμασταν αρμόδιοι είτε γιατί δεν είχαμε χώρο δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω πολλά περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ 30 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε εμείς το Δεκέμβριο και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Η Επιτροπή τώρα για το επόμενο θέμα έχει λίγα λεπτά στη διάθεσή της για να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή. Κύριε Ελκρενιέ, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένοι από εσά θα θυμόσαστε ότι το 2007 όταν διαπραγματευτήκαμε για την οδηγία όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το θέμα της επανεπεξεργασίας τους συζητήθηκε μετά από αίτημα ορισμένων μελών της Επιτροπής σας. Εκείνη την εποχή δεν μπορέσαμε να βρούμε μία λύση γρήγορα σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Στο κείμενο λοιπόν της οδηγίας ζητούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση το αργότερο στις 5 Ιανουαρίου του 2006, ε, ε, 2006 και να υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εν λόγω έκθεση έγινε σε διάφορα στάδια. Καταρχήν είχαμε διαβούλευση με του, την Επιτροπή Πυρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα το 2007. Κάτι το οποίο μας επέτρεψε να έχουμε μια εικόνα για την νομική κατάσταση που επικρατεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια συμπληρώθηκε η έκθεση αυτή. Λίγα κράτη-μέλη απαγορεύουν την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μια μια ενότητα το δέχεται στη νομοθεσία της, αλλά οι περισσότερες χώρες δεν έχουν νομοθεσία από αυτού. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ειδική νομοθεσία είναι ε, γιατί θεωρούν ότι η απουσία μέτρων σημαίνει απαγόρευση της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στη συνέχεια έγινε διαβούλευση Ιούλιο και Αύγουστο του 2008 που μας Πέτρεψε να συμπληρώσουμε και να έχουμε ένα συνθετικό κείμενο που δημοσιεύθηκε το ΜΕΤ του 2008. Το Δεκέμβριο του 2008 δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο για να καταλάβουμε καλύτερα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με το περιβάλλον και με την οικονομία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν το Μάιο του 2009. Τέλος, είχαμε την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τους κινδύνους που υπάρχουν για την ε, υγεία ήρθαμε σε διαβούλευση με την Επιτροπή αυτή για να μπορέσουμε στην έκθεσή μας να έχουμε μια στέρεα επιστημονική βάση. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν γνωμοδότησε στις 15 Απριλίου που μας πέρασε. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να μας πει κατά πόσο η, η πανεπεξεργασία αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ορίσει τον κίνδυνο αυτό και να διευκρινίσει κατά από ποιε συνθήκε και για ποια χρήση η επανεπεξεργασία ιατροκλικών προϊόντων μία χρήση ελοχεύει κινδύνου. Η έκθεση της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 27 Αυγούστου που μας πέρασε. Η έκθεση αυτή αναλύει τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την ηθική, με την υπευθυνότητα, αναλύει επίσης τις οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Γίνεται επίση μνήα στο τι γίνεται σε διεθνέ επίπεδο. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, η έκθεση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τους τρει κύριου κινδύνους που διαπιστώνονται στην πράξη από την επενεξεργασία τέτοιων προϊόντων και που εντοπίστηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή. Πρώτο πρόβλημα είναι ότι όταν έχει έρθει σε επαφή με τον ασθενή, ένα τέτοιο προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει μικροοργανισμούς, παθογενείς και να μολύνει στη συνέχεια κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει μετάδοση ιού, άρα κίνδυνο για τον ασθενή. Έπειτα, χημικά ε, υπόλοιπα μπορεί να είναι τοξικά εφόσον επαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο προϊόν. Και τέλος μπορεί να υπάρξει και τροποποίηση των ίδιων των χαρακτηριστικών φυσιολογικών και χημικών του προϊόντος με συνέπειες όσον αφορά την ε, χρήση του. Λέει η έκθεση επίσης και η Επιστημονική Επιτροπή ότι έχει εντοπίσει ένα ειδικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την μόλυνση με πρίον και ότι πρέπει να υπάρχουν μέθοδοι καθαρισμού που είναι όμως πολύ επιθετικές και που δεν ε, συστήνονται. Μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ, διακόπτη πρόεδρο. Η έκθεση, συνεχίζει εκπρόσωπο τη Επιτροπή, θίγει επίση τι ηθικέ πτυχέ και τι πτυχέ που έχουν να κάνουν με την υπευθυνότητα. Μιλά επίση για τι οικονομικέ πτυχέ και τι περιβαλλοντικέ πτυχέ. Εν κατακλείδη. Είναι δύνατον ποσοτικά να εκφράσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει από την επεξεργασία των τεχνολογικών προϊόντων μια χρήση. Τα συμβάντα που έχουν αναφερθεί είναι λίγα, αλλά δεν έχουμε μια πλήρη κοινοποίηση αυτών είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τη ζημιά που γίνεται. Δεν υπάρχει ποσοτική έκφραση όπως σας είπα. Τρεις είναι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν. Όλα τα προϊόντα αυτά δεν είναι κατάλληλα για επανεπεξεργασία και για να μειωθούν οι κίνδυνοι πρέπει να επανεκτιμηθεί όλος ο κύκλος από τη συλλογή μετά την πρώτη χρήση μέχρι την απολύμανση και την παράδοση του προϊόντος. Τώρα ποια είναι τα επόμενα στάδια μετά από την έκθεση αυτή. Αξιολογούμε τα μέτρα που θέλουμε να προτείνουμε προκειμένου να επαναχρησιμοποιούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Θα εκτιμήσουμε τις συνέπειες όλων αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ευχαριστώ, αλλά βλέπετε έχουμε και διερμηνείς που πρέπει να τελειώνουν στις 6.30 κανονικά. Οπότε λυπάμαι που σας αναγκάζω να δουλέψετε κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά τι να κάνω. Θα δώσω το λόγο για τελευταίες παρατηρήσεις στον κύριο Μέκη και στην κυρία Ροτβέρεν. Παρακαλώ. Ah, Frau vielen Dank. Hierdurch werden meine Befürchtungen bestätigt, dass also Sicherheitslücken. Υπάρχουν ε, πράγματι ε, κενά σε αυτό το σύστημα και θα θέλαμε όλα αυτά να ρυθμιστούν στο πλαίσιο ενός ε, κανονισμού. με την έννοια ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι αριθμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αρκετοί άνθρωποι πεθαίνουν από υπατήτα Β και Γ και δεν γνωρίζουμε ε, πόσοι έχουν μολυνθεί από μη καθαρή ιατρική. Ακόμα και αν είναι μικροί οι αριθμοί, νομίζω παρόλα αυτά με έναν κανονισμό μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό τους. Ε, είναι απαραίτητο επίσης να υπάρχει και υποχρέωση δήλωσης ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν ένα ε, προϊόν να επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε μία χώρα και για μία μόνο φορά και σε άλλο κράτος μάλλον να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επανειλημμένα μία πολλαπλή χρήση του προϊόντος. Πρέπει όλα αυτά να ρυθμιστούν. Η Συμφωνώ 100% ε, με τον κύριο Ούλμαρ. Η ε, παλιά νομοθεσία για τα ε, ιατρικά εξαρτήματα είναι απαρχαιωμένη. Χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη, ένα ξεκάθαρο κανονισμό. Η κυρία Μαλιόρη, πρώην Ευρωβουλευτής, προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε την πολλαπλή χρήση πρέπει ε, να την απαγορεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν ο κατασκευαστής ε, να κρίνει μόνος του που θα πουλήσει το προϊόν του. Και single use δεν σημαίνει ε, στον ίδιο ασθενή για τρεις εβδομάδες, αλλά μία και μόνο φορά. Και εάν θέλουμε η μία και μοναδική χρήση να ισχύει αυτό, εάν υπάρχει επαναχρησιμοποίηση, κάτι που κάνουν όλα τα νοσοκομεία στην Ευρώπη, είτε θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε αυτό το θέμα, είτε να θεσπίσουμε αυστηρότερους κανονισμούς. Και αυτό το χρειαζόμαστε επιγόντως. Αρχές του 2012 είναι το αργότερο που ελπίζω ότι θα αρχίσει να ισχύει αυτός ο κανονισμός. Αγαπητοί συνέδελφοι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ζητώ συγγνώμη που ήταν όλα εσπεσμένα τώρα στο τέλο. αλλά δεν είχαμε χρόνο στη διάθεσή μας. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε στις 10 η ώρα.